Well, Καλώς ήρθατε όλοι. Καλή, καλά καταφέραμε να έχουμε αυτή τη συνεδρίαση για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης ε, τη 17η. Έχουμε διερμηνία στα αγγλικά, ελληνικά, στη γλώσσα του Μαυροβουνίου. Μπορείτε να μιλήσετε γαλλικά και ιταλικά ε, Έχουμε λοιπόν διερμηνία από γαλλικά και ιταλικά, όπως και το μεσημέρι. Καλώς ορίζω και τις δύο αντιπροσωπείς, κυρίως τους συναδέφους από το Μαυροβούνιο. Κάποιοι από αυτούς έφτασαν χθες και κάποιοι άλλοι μόλις πριν από λίγες ώρες. Χαίρομαι που τα κατάφεραν όλοι να καταφτάσουν ασφαλείς. Καλωσορίζω τους συγκεκριμένους τον συμπρόεδρο και συνάδελφο, Άιβαν Μπράιοβιτς, πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου και συμπρόεδρος της Επιτροπής. Είναι χαρά που συνεργαζόμαστε για μία ακόμη φορά. Ο κ. Αλεξάνδρ Τζέζοβικ, επικεφαλής διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μιλήσει εκ μέρους της κυβερνήσεως του Μαυροβουνίου. Η κυρία Καμπριέλα Τσότ, η κυρία Τσότ είναι υπουργό για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις για τη Ρουμανική Προεδρία και ο Τόμας, επικεφαλής της μονάδας για το Μαυροβούνιο στη Γενική Διεύθυνση για την ε, Διεύρυνση και την ε, Γειτονία, τα μίση εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Μόρα Κλούν, πρόεδρος του ε, Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, που θα μιλήσει εκ μέρους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ όλους. Το εκτιμούμε ότι καταφέρατε να έρθετε. Θα ήθελα να πω κάποια λόγια εν είδη πριν μπούμε στα σημεία της ημερήσιας διάταξης και πριν ακούσουμε τους φιλοξενούμενούς μας. Καταρχάς, δεν χρειάζεται να το πω, αλλά είναι σημαντικό να τονιστεί παρ' αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να υποστηρίζει ενεργά τις επαφές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με το Μαυροβούνιο εν ώψη ε, Το βλέπουμε σαν έναν τρόπο που εξασφαλίζουμε συνεχή ανάπτυξη και ευημερία της χώρας και θεωρούμε ότι η δουλειά που κάνουμε εδώ στην Επιτροπή μας είναι πολύ σημαντική συνεισφορά στην όλη διαδικασία. Όπως ξέρετε, αυτή θα είναι η τελευταία συνεδρίασή μας κατά διάρκεια αυτής της θητείας. Από το 2014 μέχρι το 2019 ήταν η διαξετία, θα γίνουν ευρωεκλογέ από 23 μέχρι 26 Μαΐου. Οπότε και αυτή θα είναι η τελευταία συνεδρίασή μου ως συμπρόεδρος, να ευχαριστήσω ξανά τον συμπρόεδρο και τους αντιπροσώπους του Μαυροβουνίου και τους συναδέλφους του Ευρωκοινοβουλίου για την υποστήριξή τους στο ρόλο αυτό και την ενεργό συμμετοχή τους στην αντιπροσωπία. Σημειώσεις μου, κάτι λένε για το Brexit, αλλά θα έχουμε τόσο πώς εξελίξει στο Brexit που δεν θα τα αγγίξω καν αυτό το θέμα τώρα. Θα γνωρίσουν συνάδελφοι, το Ευρωκοινοβούλιο θέτησε ένα ψήφισμα για την έξι Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Μαυροβούνιο στην Ολομέλεια πέρσι. Ο Τσάρλ Τάνοκ ήταν εισηγητή, δεν έφτασε ακόμα. Μου είπε όμω ότι πρόκειται να καταφτάσει, αλλά παραμένει αυτή η οριστική θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τι τις διαπραγματεύσει. διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να συγχαρώ του συναδέλφου από το Μαυροβούνιο για τη σημαντική πρόοδο που επετεύχθη όσον αφορά τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει στου λίγου μήνε που πέρασαν από την προηγούμενη συνεδρίαση. Δεν θα αναφερθώ σε όλα τα κεφάλαια. Θα τα ακούσουμε αυτά από του άλλου φιλοξενούμενου μα, εκπροσώπου τη κυβερνήσεω, τη Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πω ότι το Μαυροβούνιο ήδη βλέπει το φω στο τέλο του τούνελ. Έχει ανοίξει σχεδόν όλα τα κεφάλαια και η γενική προτεραιότητα για το Μαυροβούνιο θα έπρεπε να είναι τώρα να εστιαστεί επιπληρώσεω των εσωτερικών κανόνων για το κράτος δικαίου, κεφάλαια 23 και 24 και μετά τη συνεδρίασή μας κάποια, κάποια άλλα πρότυπα σε άλλα κεφάλαια που θα πρέπει να τα πετύχει. Το να ανοίγει κανείς τα κεφάλαια είναι καλό, το να τα κλείνει κανείς είναι ακόμα καλύτερο και αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Πέρα από το κράτος δικαίου, που θα είναι πολύ βασικό για να κλείσουν τα κεφάλαια για μας το Ευρωκοινοβούλιο, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και θα ήθελα να πω επί τη ευκαιρία ότι εκτιμώ το ότι οι αρχές του Μαυροβουνίου έκανε σημαντικό βήμα ρίχνοντας φως στην επίθεση κατά της Ολίβια Λάκικ, της δημοσιογράφου, που πυροβολήθηκε στο στην πρωτεύουσα στις 18 Μαΐου. Εννέα άτομα από ό,τι γνωρίζουμε μέλη εγκληματική οργανώσεω συνελήφθησαν τον περασμένο μήνα και συνδέονταν με αυτό το εγκλήμα και καλωσορίζω τι μέχρι τούδε καταβληθεί προσπάθειε για την εξυχνίαση αυτού του αποτροπιαστικού εγκλήματο. Και καλούμε τι αρχέ του Μαυροβουνίου να συνεχίσουν τι έρευνε μέχρι ότου να ρηχθεί άπλετο φω στην επίθεση, κίνητρα και όλοι οι εμπλεκόμενοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Η ελεύθερα μέσα ενημέρωση είναι ακρογωνιαίο λίθο δημοκρατική κοινωνία και θα πρέπει να μην υπάρχει ατιμορρησία για τέτοιε επιθέσει κατά δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να μπορούν να ζουν σε ασφαλέ περιβάλλον χωρί να φοβούνται δίωξη, να είναι προστατευμένοι από το νομοθετικό πλαίσιο. Και σχετικά με αυτό, καλωσορίζω τη δέσμευση του Μαυροβουνίου να ακολουθήσει τι βέλτιστε πρακτικέ και να αρμονίσει την νομοθεσία του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεκτημένο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, να τονίσω κάτι πάνω από πέντε χρόνια μετά την, το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24, η γενική πρόοδος όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης παραμένει κάτι που δεν είναι ικανοποιητικό και προειδοποιώ, όπως λέει και η έκθεση, κατά εσδήποτε πολιτικής παρεμβολής στο έργο των εθνικών δημοσίων εταιριών μέσων του κυβερνήσεως, του κρατικών, και δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τη διάθεση ε, δημοσίων πόρων στα μέσα στη, στο Μαυροβούνιο και θα πρέπει οι αρχέ να θετήσουν την κατάλληλη νομοθεσία τους ώστε να εξασφαλίζουν την ποικιλομορφία και τη βιωσιμότητα των μέσων ενημέρωση. Σχετικά με την παρούσα κατάσταση για τι σοβαρέ κατηγορίε για ε, διαφθορά και παράνομη χρηματοδότηση των κομμάτων, θετική εξέλιξη είναι η έκτακτη σύνοδο όσον αφορά την υπόθεση για φακελάκια που έγινε στι 21 Φεβρουαρίου είναι πολύ σημαντικό τώρα οι αρμόδιες αρχές και οι θεσμοί να δράσουν γρήγορα και αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσουν αυτές τις κατηγορίες με έναν τρόπο ανεξάρτητο. Όσον αφορά τη συνεχ... τη συνεχή, το συνεχέ μποϊκοτάζ των εργασιών του Κοινοβουλίου από πλευρά τη αντιπολιτευσίω, εγώ είμαι απογοητευμένο που βλέπω ότι για δεύτερη φορά έχουμε μόνο ένα κόμμα τη αντιπολιτεύσεω που εκπροσωπείται εδώ. Τούτου λεχθέντο χαίρομαι που ο κ. Κρυβάκοπιτ μπόρεσε να έρθει εδώ, τον ευχαριστώ. Η θέση μας σχετικά με αυτό παραμένει αμετάβλητη. Όλη η αντιπολίτευση θα πρέπει να επανέλθει στο Κοινοβούλιο, διότι εκεί θα πρέπει να διεξάγεται η πολιτική συζήτηση. Ο πολιτικός διάλογος είναι βασικό στοιχείο δημοκρατικού συστήματος και βασικό βήμα συζητήσεων θα πρέπει να είναι το Κοινοβούλιο που λειτουργεί πλήρω. Πιο σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτό, μέσω των υποθέσεων που ξέσπασαν όσον αφορά τα, τις δωροδοκίες, τα φακελάκια κλπ. Εξού σημαντικό θα είναι η Επιτροπή του Κοινοβουλίου για την εκλογική μεταρρύθμιση να καταλήξει στο να πετύχει τους στόχους της φιλόδοξης ατζέντα της. Σχετικά τώρα με τη διαμαρτυρία που συνεχίζεται, αυτή, έτσι λειτουργεί η κοινωνία δημοκρατική, η κινητοποίηση των πολιτών είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Είναι κρίσιμο λοιπόν η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου θα πρέπει να ε, καλύψει τι ανησυχίε των πολιτών. Και τέλο, κάτι εξίσου σημαντικό, από 23 μέχρι 26 Μαου θα έχουμε τι εκλογέ για το Ευρωκοινοβούλιο και πιστεύω και ελπίζω ότι το επόμενο Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να υποστηρίζει διεύρυνση, την πολιτική διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεπώ την ένταξη του Μαυροβουνίου που είναι στην πρώτη γραμμή τη διαδικασία. Ελπίζω ότι μέχρι να γίνουν εκλογέ του 2024 να συμμετέχουν οι Μαυροβούνιοι σε αυτές τις ε, εκλογέ. Βέβαια, εξαρτάται αυτό από τη συνέχιση της ουσιαστική προόδου και στο κλείσιμο των εναπομενών των κεφαλαίων. Πολλά από αυτά τα σημεία θα τα έχουμε στην ημέρησια διαταξή μα, αλλά πριν προχωρήσουμε και πάμε στην ημερήσια διάταξη αυτή κάθε αυτή. Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντα το λόγο στου διάφορου φιλοξενούμενου μα να μιλήσουν για το πώ πάνε οι διαπραγματεύσει και καταρχά να δώσω το λόγο στον επικεφαλή των διαπραγματεύσεων, ώστε θα μπορέσει. Α, συγγνώμη, στον συμπρόεδρο πρώτα. Στον συμπρόεδρο πρώτα να του δώσω το λόγο. Hvala. Καλησπέρα σα. Συμπρόεδρε Μάρτιν, κυρίε και κύριοι, είμαι εδώ και με πολύ χαρά θα συζητήσω τι εξελίξει στο Μευροβούνιο καθώ και την διαδικασία σύνδεσή. Του τελευταίου τέσσερι μήνε, παρότι που συνδεθήκαμε, συνέβησαν πολλά τα οποία απαιτούν την προσοχή μα. Έχουμε εκλογές το 2020. Μετά από τις τελευταίες εκλογές η πλειοψηφία βελτιώνει το κλίμα βάσει των συστάσεων διεθνών παρατηρητών. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στις εκλογικές διαδικασίες. Για ο μιλητής. Transition. Uh, Το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου δημιούργησε μια διάμεση επιτροπή για την εκλογική διαδικασία και θέσπισε και άλλους νόμους. Στόχος όλων των κομμάτων στο Μαυροβούνιο είναι αυτός. Ο διάλογος είναι η μόνη προσέγγιση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αποδεκτό αποτέλεσμα για όλους τους εμπλεκομένους στην πολιτική ζωή του Μαυροβουνίου. Προσπαθούμε επίσης να βελτιώσουμε τις συνδίκες του κράτους δικαίου. Κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης το έπραξαν και αυτά, αλλά μάλλον προσχηματικά. Θα προτιμούσαν να μην γίνει κανένας διάλογος Και το διότι υπεραμείνονται διαφόρων ε, δομών και προσεγγίσεων που δεν μπορούν να αποτελούν μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Νομίζω ότι γι' αυτό επέλεξε να μην συμμετέχουν στις εκλογές έως ότου τα πράγματα γίνουν όπως τα θέλουν. Και αυτό δυστυχώς δεν βαίνει προς την ομοιοποίηση των δημοκρατικών μας θεσμών. Φοβούμαι ότι η αντιπολίτευση καταχράτε των δημοκρατικών θεσμών. Και συνεχίζουν να ισχυρίζονται και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. λοιπόν, αβάσιμα επιχειρήματα. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι ως μέλος του ΝΑΤΟ και ως χώρα η οποία έχει ευρωπαϊκές φιλοδοξίες, στόχος μας είναι να έχουμε διάλογο μεταξύ θεσμών στον Μαυροβούνιο δεν γίνεται να ενισχύσουμε το κράτος μας, να το σταθεροποιήσουμε, εάν δεν εξασφαλίσουμε διάλογο. Τονίζω λοιπόν τον ρόλο των μέσων προκειμένου. Την ανάγκη μια επαγγελματικής προσέγγισης. Δεν μπορεί κανείς να αξιοποιεί, να εκμεταλλεύεται αβάσιμες πληροφορίες και ισχυρισμού για ιδίου σκοπούς. Ορισμένοι υποτιμούν το αποτέλεσμα των ίδιων των εκλογών φοβούμε, ότι δημιουργούν τεχνιέντος θόρυβο για να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Σε τέλη του Φεβρουαρίου η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δρομολόγησε μια έκτακτη σύνοδο του Κοινοβουλίου. Είχαμε συζήτηση επί ισχυρισμών περί διαφθοράς, παρανομής χρηματοδότησης κομμάτων κλπ. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία πιστεύει ότι ο διάλογος πρέπει να γίνεται στη Βουλή. Ανέκαθεν υποστηρίξαμε ότι δεν θα γίνουμε θύματα, δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς. Πιστεύω ότι οι ρεαλιστικές απόψεις θα επικρατήσουν, οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις θα επικρατήσουν και ότι θα συνεχίσουμε στον δρόμο της πλήρους ένταξης. Θέλουμε να ανοίξουμε και τα τελευταία κεφάλαια και φυσικά να αρχίσουμε να κλείνουμε κεφάλαια οριστικά. Η εντολή της Επιτροπής μας, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, είναι βεβαίω να συνεχίσουμε στον δρόμο της διεύρυνσης τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τα Βαλκάνια, κάτι το οποίο θα είναι προ όφελο τη σταθερότητα. Εύχομαι σε όλου μια επιτυχή σύσκεψη σήμερα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίηση και Σύνδεση. Ευχαριστώ πραγματικά για όλα όσα κάνατε ω σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Θεωρώ ότι ενεκρίθη η ημερήσια διάταξη. Για τα περασμένα πρακτικά δεν υπάρχει κάποια αντιρρήση φαντάζομαι. Περνάμε στο υπερθυμό 3. Εξέλιξη των ε, ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ε, τον λόγο στον επικεφαλής διαπραγματευτή από την πλευρά του Μαυροβουνίου. Κυρίε και κύριοι, καλώ ήλθατε. Κύριε Πρόεδρε, Μάρτιν και Μπράγιοβιτς μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Είναι μεγάλη η χαρά μου που είμαι εδώ σήμερα και που έχω τη δυνατότητα να σας παρουσιάζω τις πιο σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά τη διαπραγματεύση για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι προχωρούμε σε συνεργασία με τη Βουλή και τη συνένεση όλων των κομμάτων στον δρόμο της ένταξης. Η συνέντευξη αυτή, ξέρετε, είναι σπάνια. Αλλά αυτό αποτελεί και ένα επιπλέον κίνητρο να ολοκληρώσουμε το έργο μας το συντομότερο δυνατόν. Υπολογίζουμε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο ανέκαθεν υπεραμείνθηκε τη ευρωπαϊκής μας προοπτικής. Και το λέω αυτό διότι διστάμενες απόψεις ακούστηκαν από κάποια κρατημέλη. Όσον αφορά τώρα τις διαπραγματεύσεις, το 2018 ανοίξαμε τα κεφάλαια, 26, 27 με συγχωρείτε, είναι το 32ο κατά σειράν, οπότε τα μη ανοιγμένα κεφάλαια δεν είναι παρά ένα, το 8, ανταγωνισμός. Η θέση που ενέκρινε και η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου είναι ότι έχουμε ολοκληρώσει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, οπότε με το που θα κληθούμε μπορούμε να παρουσιάσουμε και την σχετική διαπραγματευτική μας θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε ότι η κατάρτιση των διαπραγματευτικών θέσεων δεν θα πάρει χρόνο για να μπορέσουμε, όπως προείπα, να ανοίξει και το τελευταίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της Ρουμανικής Προεδρίας. Προχωρούμε λοιπόν πολύ ικανοποιητικά, θεωρώ, στην υλοποίηση και των ειδικών μας υποχρεώσεων. Κάθε κλείσιμο κεφαλαίου είναι και αναγνώριση των προσπαθειών της κυβέρνησης και της διοίκησης και αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πορεία ένταξης. Σκοπεύουμε να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπαθειές μας, να τις επιταχύνουμε μάλιστα, στο χέρι μας είναι άλλωστε, αλλά περιμένουμε το ίδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα και την κοινή γνώμη. Να υπογραμμίσω ότι η υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική για μα. Για να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, με την ίδια ταχύτητα, με την ίδια ορμή, εμεί ε, δεσμευόμαστε να τηρήσουμε τους ενδιαμέσους σταθμούς. Το Μαυροβούνιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να χάσουν χρόνο θα ήταν κρίμα μετά από τα όσα έχουμε πετύχει. Μέχρι στιγμής πάντως, παίρνουμε βάση χρονοδιαγράμματος. Έχουμε τώρα το κεφάλαιο 23 και το 24. Τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και αυτά εξέλιξονται όπως είπα κανονικά. Ήδη υλοποιούμε και ένα μεγάλο κομμάτι του 23 και του 24 και είμαστε στο 75% όσον αφορά το κεφάλαιο 24. Όλα αυτά αποδεικνύουν ακριβώς την ε, δέσμευσή μας στην διαπραγματευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό, το Μαυροβούνιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην ελευθερία των μέσων και στην ελευθερία της έκφρασης. Ήδη προετοιμάζουμε νέο νόμο για τα μέσα και νέο νόμο για την κρατική ραδιοτηλεόραση. Θα έτσι τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελευταία της άτυπη ανάλυση του τομέα στο Μαυροβούνιο διαπιστώνει συνεχή βελτίωση στις νομοθετικές διαδικασίες, στη δημιουργία θεσμών καθώς και στα πρώτα αποτελέσματα του αγώνα για την πάταξη της διαφθοράς, του ξεπλήματος, μαύρου χρήματος και την δίμευση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Μάλιστα, η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια, χάρη ακριβώ στην καλύτερη αστυνομική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι εθνικέ αστυνομίε. Είμαι πεπισμένο ότι η συνεργασία αυτή κατά του οργανωμένου εγκλήματο αποτελέσει μια ισχυρή βάση για τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι αυτά θα αποτυπωθούν και στις μελλοντικέ εκθέσεις. Όλα αυτά θα μας φέρουν ακόμη πιο κοντά για να μπορέσουμε για να μπορέσει μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βεβαιώσει ότι έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Και στο επόμενο στάδιο, στάδιο με συγχωρείτε, θα κλείσουμε και τα κεφάλαια που αφορούν το κράτος δικαίου πολύ σημαντικό για τι ενταξιακές διαπραγματεύσει. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, έχουμε ήδη εκπληρώσει όλε τι υποχρεώσει μα για να κλείσουν και άλλα κεφάλαια. Τα περισσότερα λοιπόν θεωρώ το έχουμε κάνει στο κεφάλαιο 6 για παράδειγμα, στο 7 πνευματικά δικαιώματα, στο 10 πληροφορική και τεχνολογία, στο 21 διευρυπαϊκά δίκτυα και στο 30. Ένα για την εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Εν προκειμένου το Μαυροβούνιο δεσμεύεται επίση να τροποποιήσει την διαδικασία για να ενσωματωθεί, να εναρμονιστεί μάλλον με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Όσον αφορά την ποιότητα αυτή τη διαδικασία, υιοθετούμε κανονισμού. Η Κομισιόν επιμένει επ' αυτού, το καταλαβαίνουμε, για να μπορέσουν να κλείσουν και άλλα κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η εφαρμογή να γίνει στην πράξη. Εδώ χρειάζεται λίγο περισσότερος χρόνος. Αλλά θα γίνει και αυτό σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Μαυροβούνιο. Το θέμα είναι να θέσουμε ρεαλιστικές προθεσμίες για την εφαρμογή στην πράξη της νομοθεσίας. Το ίδιο ισχύει και για την μεταρρύθμιση των θεσμών και την δημιουργία ικανοτήτων, όπως ε, λέγεται. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο πρέπει να υποστεί πολλές αλλαγές για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην ένταξη. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει στηρίξει, αλλά και πολλά κράτη-μέλη μας έχουν στηρίξει, τα οποία μας παρέχουν πολύτιμη βοήθεια. Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, το Μαυροβούνιο πέτυχε σημαντική ταχεία, ταχύ οικονομική ανάπτυξη, θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο της δημοσιονομικής εξηγένσης. Το 2019 εκτιμούμε ότι θα είναι το έτος της πρώτης μείωσης του ελλείμματος του προπολογισμού. Το Μαυροβούνιο παραμένει προσιλωμένο στον δρόμο της Ευρώπης, αλλά και στην βελτίωση των καλών σχέσεων γειτονία με χώρες με τις οποίες συμμεριζόμαστε κοινέ αξίες. Το Μαυροβούνιο, κυρίε και κύριοι, βαδίζει στον δρόμο της Ευρώπη, όπω είπα, το όραμά μας είναι σαφέστατο. Θέλουμε μια καλύτερη κοινωνία. Θέλουμε να αναπτυχθούμε ως σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων πιστεύω ότι σημειώσαμε ορατή, απτή πρόοδο και αυτό θα είναι και μια καλή βάση για τις μελλοντικέ εξελίξει. Η βούληση υπάρχει, έχουμε τη βούληση να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις και θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω ότι αυτό θα συνεχίσει να ισχύει και στο μέλλον. Από την άποψη αυτή και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τις ευκαιρίες που μας δώσατε, για την υποστήριξή σας. Χαίρομαι πραγματικά που προχωρούμε στον δρόμο της ένταξη. Αυτό ήταν προτεραιότητα και της προηγούμενης Προεδρίας, αλλά και της Ρουμανικής Προεδρίας. Ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει και η επόμενη εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωση Έτσι αυτή η πολύ σημαντική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηριχθεί και από, την επόμενη, και από το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας στραφούμε τώρα. Προς την κυρία Τσότ. Εντάξει, το είπα σωστά. Κυρία Τσότ, που είναι υπουργό για θέματα Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, και εκπροσωπεί τη Ρουμανική Προεδρία. Αγαπητή συμπρόεδρε, επικεφαλή των διαπραγματευτών, αξιότιμα μέλη, κυρίε και κύριοι, εκ μέρου τη Προεδρία ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είναι μεγάλη χαρά να μπορώ να σα απευθύνω τον λόγο επί τη ευκαιρία αυτή τη 17η συνεδριάσεω Τη κοινοβουλευτική επιτροπή για σύνδεση και σταθεροποίηση του Μαυροβουνίου. Ευπρόσδεκτος επικοδομητικό ρόλος αυτή τη Επιτροπής για την ενταξιακή διαδικασία του Μαυροβουνίου και εν γέννη το Ευρωπαϊ... καλωσορίζουμε και την σταθερή υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου για την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα ξέρετε σίγουρα ότι η Ρουμανική Προεδρία εν γέννη θέλει να εφαρμόσει αυτή την πολιτική διότι πιστεύουμε ότι είναι το αποτελεσματικότερο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την εξασφάλιση ειρήνης, δημοκρατίας, ευημερίας και σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης μέσω μεταμορφωτικής δυνάμεως και σαφών ωφελών που δίδει στους πολίτες. Τώρα, όσον αφορά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο, που άνοιξαν σχεδόν πριν από 7 χρόνια και θέλουμε να προωθήσουμε ευπρόσδεκτη το καθεστώς σας ότι είσαστε στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την δεξιακή διαδικασία και συγχαρητήρια και την επιτευχθήσα πρόοδο τελευταίο έτος. Αυτό αποδεικνύεται από ότι σχεδόν όλα τα κεφάλαια έχουν ανοίξει. Σαν αξιόπιστο εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ενώσης στην περιοχή, το Μαυροβούνιο παίζει θετικό και επικοδομητικό ρόλο για την πρόθεση περιφερειακής συνεργασίας και των καλών γειτονικών σχέσεων. Και πενούμε τη συνεχή συνεργασία του Μαυροβουνίου για θέματα εξωτερικής πολιτικής και την πλήρη ευθυγράμμιση αυτού με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμεσα Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ταυτόχρονα είναι σαφές ότι η παρούσα κατάσταση είναι πολύ απαιτητική. Έκανε προσπάθειες στο Μαυροβούνιο πάνω σε διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εγκρίσεως ε, σημαντικών μέσων στον τομέα του κράτους δικαίου και δημιουργήθηκαν διάφοροι θεσμοί. Παρ' όλα αυτά το Μαυροβούνιο δεν μπόρεσε να ε, οδηγήσει κεφάλαια σε προσωρινό ε, κλείσιμο. Για να προθεθεί διαδικασία θα πρέπει να δώσει απτά αποτελέσματα το Μαυροβούνιο, κυρίως στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της καταπολεμήσεως της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, του ξεπλήματος χρήματος και του εμπορίου ε, σαρκός, εμπορίου ανθρώπων και θα πρέπει να προωθήσει την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης. Η κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει ισχυρή πολιτική βούληση για εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών. Θα πρέπει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσει που έχει αναλάβει και να πετύχει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα. Τέτοια βιώσιμη πρόοδο θα επιτρέψει το κλείσιμο και άλλων κεφαλαίων οι ανησυχητικέ επιθέσει κατά δημοσιογράφων που έγιναν πέρσι και εξελίξει όσον αφορά τι δημόσιε το RTCG, τον κρατικό σταθμό και την υπηρεσία για τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, δείχνει τη σημασία που έχει να εγγυηθούν ασφαλές κλίμα για τα μέσα ή αρχές, όπου εκεί να μπορούν οι δημοσιογράφοι να ασκούν ελεύθερα το επάγγελμά του. Άλλο στόχο πρέπει να πετύχει το Μαυροβούνιο είναι συνεχείς προσπάθειες για διοικητικό δυναμικό σταθερό και περισσότερη τεχνογνωσία πρέπει να αποκτηθεί για τον πολιτικό διάλογο. Έληξε ο μακροσκελής πολιτικός κύκλος των εκλογών και όλοι οι φορείς οι πολιτικοί θα πρέπει να συνεργαστούν επικοδομητικά και μεταξύ τους και με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις αυτής για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα μελλοντικά που θα εμφανιστούν με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται περισσότερες προσπάθειε για να γίνει μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου, ούτω ώστε διαδικασία να καλύπτει όλου και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη όσον αφορά το εκλογικό πλαίσιο. Αυτέ οι προσπάθειε, αν γίνουν, μπορούν να ανανεώσουν την όλη όθηση που θα έχει πορεία του Μαυροβουνίου προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να ανοίξει το κεφάλαιο 27 για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματο στην τελευταία κυβερνητική το Δεκέμβριο έδειξε ότι το Μαυροβούνιο μπαίνει στην επόμενη φάση της ενταξιακής διαδικασίας Εκεί αναμένεται να εστιαστείτε επιλοπίσεως μεταρρυθμίσεων με αποφασιστικότητα και να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι. Τα, τα υπόλοιπα που πρέπει να ανοίξουν και αυτά πρέπει να κλείσουν τα κεφάλαια και τα ενδιάμεσα κεφάλαια, όπως και το 23 και 24 πρέπει να προωθηθούν. Όπως είπε και το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του του περασμένου Ιουνίου, σαφής πρόοδος και πραγματικά αυτά αποτελέσματα όσον αφορά το κράτος δικαίου είναι ο αποσυστικός παράγοντας για τη γενική βάση των διαπραγματεύσεων. Εμείς ενθαρρύνουμε το Μαυροβούνιο να δράξει αυτή την ευκαιρία και να συνεχίσει να εφαρμόζει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις υπό το φως της εκθέσεως του 2018 για το Μαυροβούνιο και βάσει των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Ιουνίου 2018, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και την επικείμενη το ετήσιο πακέτο για τη διεύρυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έκθεση πρόοδου αυτής. Σας διαβεβαιώνω και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη και η Ρουμανία σαν προεδρεύουσα του Συμβουλίου ένθερμα θα υποστηρίζουμε ε, το Μαυροβούνιο στη διαδικασία μεταρρυθμίσεως. Κλείνοντας, καλωσορίζω τι προσπάθειε που καταβάλει η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για να προωθήσει την ενταξιακή διαδικασία και αυτό δίνει μια υπόσχεση για καλύτερο μέλλον και για του πολίτε και για τη χώρα, η ένταξη. Εμεί, η Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, ε, σα διαβεβαιώνουμε και ότι και η διεύρυνση και τα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθούν να έχουν ψηλή θέση στο θεματολόγιο μας. Α, υπό τον όρο ότι θα πληρωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ελπίζουμε να μπορέσουμε να προεδρεύσουμε μια άλλη διασκέψεως τον Ιούνιο για να επενθυμίσουμε την πρόοδό σας και να ξεκινήσουν ε, με το άνοιγμα ε, του κεφαλαίου του τελευταίου για τις πραγματεύσεις, του κεφαλαίου 8 για τον ανταγωνισμό. Και θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί το Μαυροβούνιο να προωθεί στη διαδικασία. Καλούμε όλους τους εκπροσώπους του Μαυροβουνίου που είναι εδώ παρόντες σήμερα να αρπάξουν αυτή την πολιτική ευκαιρία να αυξήσουν τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση εδραζόμενοι επί της επιτευθύσας προόδου και να εστιαστούν επί της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικά επικοδομητικά και τώρα επικεφαλή μονάδα για το Μαυροβούνιο στη Γενική Διεύθυνση Γειτονία και Διεύρυνση και Διαπραγματεύσει. Ο Τόμα ήταν πάντα ε, παρόν σε αυτή την επιτροπή και εδώ και στο Μαυροβούνιο και συμμετείχε ένθερμα και στις Βρυξέλλες και ευχαριστώ Τόμας για αυτή την αφοσίωσή σου. Ευχαριστώ κύριε Μάρτιν, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, όπω ο κύριος Στέλεβη και ο κύριο Κράγιοβιτ είπαν, θα ήθελα καταρχάς και εγώ να αποτίσω φόρο τιμής προς τον συμπρόεδρο μας, τον κύριο Μάρτιν, και τη συνεισφορά τους ε, στο έργο αυτής της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, Σταθεροποίησης και Ένταξης. Αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια που καταβάλατε. Ήταν σημαντικό χρήσιμο στοιχείο στο διάλογο μεταξύ των κοινοβουλίων. Ξεκινώντας, θέλω να επενθυμίσω τη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετήθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου και σαφώς επιβεβαιώνει τις προοπτικές που έχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων συμπεριλαμβανομένου του Μαυροβουνίου και ανακοινώθηκε ότι θα αυξηθεί η προσπάθεια και οι επαφέ Ευρωπαϊκή Ένωση με όλη την περιοχή. Και η στατική επιβεβαιώθηκε και στη Σύνοδο Κορυφή στη Σόφια, στη διακήρυξη τη Σόφια, και στην ατζέντα της Σόφιας και από τον Ιούνιο του Συμβουλίου, όλα αυτά θέτουν το πλαίσιο εντός του οποίου και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κινηθεί όσον αφορά την ενταξιακή διαδικασία και ένα σαφές μήνυμα ενθάρρυνσης για την ενταξιακή διαδικασία του Μαυροβουνίου καθώς και για τους γείτονες του Μαυροβουνίου. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το Μαυροβούνιο, να πω μερικά λόγια για την πολιτική κατάσταση και για την ενταξιακή διαδικασία που βρίσκεται. Όσον αφορά την πολιτική κατάσταση, ο πολιτικός διάλογος νομίζω παραμένει βασικό στοιχείο στη χώρα και βασική μέρημνα για μας και αποτελούσε και προτεραιότητα της επισκέψης του Επιτρόπου Χάν που έγινε πρόσφατα στο Μαυροβούνιο. Πάντα υπήρξαμε σαφείς ότι ένα πλήρως λειτουργών κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό. Ο πολιτικός διάλογος ανήκει στο κοινοβούλιο. Σχετικά με αυτό καλωσορίσαμε τη σύσταση της Προσωρινής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για εκλογική μεταρρύθμιση το περασμένο φθινόπωρο. Ακόμα περιμένουμε αυτή η Προσωρινή Επιτροπή να πετύχει τους στόχους της, βελτιώνοντας το γενικό περιβάλλον διεξαγωγής των εκλογών βάσει εκθέσεω και των συστάσεων τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είδαμε απτή πρόοδο μέχρι τώρα όσον αφορά τις εργασίες αυτής της Επιτροπής. Όμως, οι παρούσες εξελίξεις επεσκίασαν το έργο της προσωρινής Επιτροπής. Αυτό δεν θα πρέπει να αποσπάσει την προσοχή μας από τη σημασία που έχει το έργο της προσωρινής επιτροπής που ανέλαβε αυτό το ρόλο και έχει σημαντική εντολή. Είδαμε πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα, αναφέρονται σαν υποθέσεις άτλας και φάκελος, θα συζητηθούν εκτενέστερα, πιστεύω αυτά. Πώς βλέπουμε τις εξελίξεις θεωρούμε ότι το Μαυροβούνιο έχει νομοθετικό πλαίσιο. Έχει τους θεσμούς για την αντιμετώπιση αυτών των κατηγοριών που εμφανίστηκαν. Εξατάται από τους θεσμούς η κατάσταση, όπως από τον ειδικό εισαγγελέα και τον φορέα πολεμήσεως της διαφθοράς να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταγγελίες με ανεξάρτητο και επαγγελματικό τρόπο σύμφωνα με την ανατεθήσα εντολή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία της μεταρρύθμισης για το κράτος δικαίου του Μαυροβούνιου και για την αξιοπιστία των, του θεσμικού και οικονομικού του συστήματος. Να πω κάτι όσον αφορά την ενταξιακή διαδικασία και τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Ήδη αναφέρθηκε ότι το Μαυροβούνιο είναι η πιο προχωρημένη χώρα όσον αφορά τη διαδικασία και βασικά εστιαζόμεθα επί της πληρώσεως των προσωρινών κριτηρίων όσον αφορά το κράτος δικαίου και τα σχετικά κεφάλαια η αξιολόγησή μας ακολουθεί τον συνεχή διάλογο με τις αρχές του Μαυροβουνίου. Στενότατη συνεργασία με το Μαυροβούνιο έχουμε. Είδαμε πράγματι ένα, αρχικές επιτυχίες σε διάφορους τομείς, όπως κατά οργανωμένου εγκλήματος, διαφθορά υψηλού μεγάλου επίπεδου, εξυχνίαση ξεπλήματο χρήματο, προσωπικο πάγωμα στοιχείων ενεργητικού. Πιο περιορισμένα αποτελέσματα έχουμε σε άλλου τομεί, όπω την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Είδαν περισσότερα αποτελέσματα κυρίω μέσω διεθνού ε, διευρυμένη διεθνού συνεργασία. Άλλοι τομεί, όπω η ελευθερία των μέσων όμω, οι επιθέσει κατά των δημοσιογράφων, η ανεξαρτησία των δημοσίων σταθμών, των κρατικών σταθμών, η καταπολέμηση της διαφθοράς, το εμπόριο ανθρώπων, και η κατάσχεση ε, οικονομικών στοιχείων ενεργητικού εκεί είναι τομείς που μπορούν τα αποτελέσματα να βελτιωθούν, ούτω ώστε να ανταποκριθούν στα προσωρινά κριτήρια. Τώρα όσον αφορά το εναπομένων κεφάλαιο για να ανοιχθεί το 8, σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάναμε πρόταση προς το Συμβούλιο. Συστήσαμε, είπαμε μάλλον ότι έχουν πληρωθεί τα κριτήρια για να ανοίξει το κεφάλαιο. Γίνονται συζητήσεις μεταξύ κρατών μελών επ' αυτού και προσβλέπουμε στο άνοιγμα του κεφαλαίου το ταχύτερο δυνατόν. Και μετά θα υπάρξουν προσανατολισμοί μέσω των περαιτέρω κριτηρίων που θα θεσπιστούν για να κλείσει το κεφάλαιο. Και αφορά και τη λειτουργία της οικονομίας. Τέλος. Μερικά λόγια να πω για βασικά στοιχεία της ενταξιακή διαδικασία μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκηση που γίνεται πολλή δουλειά από τι τιμή στι προσπάθειε που έγιναν μεταρρυθμίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο στόχος η ενίσχυση του επαγγελματισμού των δημοσίων υπαλλήλων Χρειάζονται καλύτερα αποτελέσματα από τη δημόσια δίκηση. Χρειάζεται βελτιστοποίηση τη δημόσιας δίκηση στο Μαυροβούνιο. Να χρησιμοποιούνται σωστά οι πόροι. Συνεργαζόμαστε με τις αρχές για να τις βοηθήσουμε να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Μαζί με την πρωταξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οικονομία, οικονομική διακυβέρνηση, Το Μαυροβούνιο έχει σημαντική οικονομική ανάπτυξη τον τελευταίο χρόνο. Ταυτόχρονα είδαμε προβλήματα με το δημόσιο χρέος, να αυξάνονται τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Παρά την σημαντική οικονομική ανάπτυξη, χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες οικονομικής εξυγίανσης στο Μαυροβούνιο και θα δώσουμε σχετικά συστάσεις για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Και εκεί θα τονίζουμε την ανάγκη για πιο ευέλικτη οικονομία, για μεγαλύτερη ποικιλομορφία στην οικονομία, βελτίωση της αγοράς εργασίας, να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να βελτιωθεί και η απασχόληση και η οικονομία. Όπως προανέφερα, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Μαυροβούνιο και μέσω τεχνικής τεχνογνωσίας και μέσω σημαντικής οικονομικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με αυτά ευχαριστώ πολύ και εύχομαι επιτυχή συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. κύριε θα μιλήσει εκ μέρους της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ για τον λόγο. Να υπενθυμίσω ότι η πρόσωπο, κύριε Μοκερίνη, έχει διατυπώσει με σαφήνεια την υποστήριξή της υπέρ της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και θα κάνει την πέραση προχέρη της προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν θα επισελθώ, δεν χρειάζεται άλλωστε στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Πάντως πέρσι πρέπει να πω ότι η προσωρινή επιτροπή για την εκλογική διαδικασία ήταν μια ευχαριστή εξέλιξη. Θα θέλαμε να δούμε ότι η επιτροπή αποδίδει όπως περιμένουμε, ότι θα δερμολογηθεί ο διάλογος και στη Βουλή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες του Μευροβουνίου, αλλά και την πρόθεση των σχετικών μεταρρυθμίσεων. Ενθαρρύνουμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα να συμμετάσχουν επικοδομητικά στον διάλογο. Παρακολουθούμε επίση από κοντά τι καταγγελίε περί ξεπλήματος βρού, χρήματο. Αυτό θα κρίνει την επιτυχία της δημοκρατίας. Οι θεσμοί, οι δημοκρατικοί θεσμοί είναι κρίσιμοι για κάθε δημοκρατία. Όσον αφορά την πολιτική ασφάλεια και άμενος, όπω είπε η κυρία Τσότ, το Μαυροβούνιο είναι ένας αξιόπιστος εταίρος, ευθυγραμμίζεται όλο και περισσότερο με τις ευρωπαϊκές θέσει. Η συνεργασία του Μαυροβουνίου σε επιχειρήσεις ειρηνευτικές και επιχειρήσεις στα θεροποίηση, στην επιχείρηση Αταλάντα μεταξύ άλλων, ήταν μεγάλη αξία. Από την τελευταία μα συνάντηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μαυροβούνιο οριστικοποίησαν σχετική συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ πολύ σύντομα όσον αφορά τις προτεραιότητες της Σόφιας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε μια διερεύνηση της κατάστασης, να δούμε ποια προγράμματα θα βοηθήσουν περισσότερο τη χώρα. Το Μαυροβούνιο λειτουργεί λοιπόν επικοδομητικότητα στον τομέα αυτών και θεωρείται ήδη ένας αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβλέπουμε σε περαιτέρω επικοδομητική συνεργασία. Τέλος, όσον αφορά το έργο του κυρίου ε, Συμπροέδρου, εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ και να περάσουμε σε συνεισφορές από τους συμμετέχοντες εν γέννη. Ο κύριος Βουξάνοβιτς, βουλευτής της ε, Βουλής του Μαυροβουνίου. Κύριε Συμπρόεδρε, κύριε Συμπρόεδρε, κύριε Μάρτιν προκειμένου. Και Μπραγιοβίτς. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Πραγματικά το κλίμα είναι εξαιρετικά επικοδομητικό και επικοδομητικά θα μιλήσω και εγώ για το βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του Μαυροβουνίου. Πρόκειται για μονόδρομο θα έλεγα για το Μαυροβούνιο να ευχαριστήσω τον κύριο Μπράγεβιτς και τον κύριο Κουτέλεβιτς, οι οποίοι υπογράμμισαν τα κύρια γεγονότα που συνέβησαν δηλαδή από την περασμένη μας συνάντηση σήμερα. Εγώ λοιπόν να πω λίγα πράγματα περισσότερα όσον αφορά την ενταξιακή μας πορεία. Πρώτον, Έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε ακριβώ χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των άλλων θεσμικών οργάνων που εμπλέκονται στην διαδικασία. Από στατιστικής απόψεως, αν θέλετε, όσον αφορά την πρόοδο που σημειώσαμε, θα έλεγα ότι στις 22 Νοεμβρίου να σας θυμίσω την τελευταία μας σύσκεψη. Ο κ. έχει λάβει μέρος. Λάβαμε υπόψη μας την ένατη έκθεση πεπραγμένων για την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου 2018. Και μετά είχαμε και την 7η τριμηνία έκθεση Μελετήσαμε επίση την εξαμηνία έκθεση, όπως είπα, Ιανουάριος-Ιούνιος, η οποία ενεκρίθη στην προηγούμενη σύνοδο της Επιτροπής μας, τον Δεκέμβριο. Το κείμενο θα μπορούσε να θεωρηθεί πληκτικό, θα έλεγα, και όμως αποτυπώνει τη δέσμευση της Βουλής του Μαυροβουνίου να συνεισφέρει ουσιοδό στη διαδικασία. Πρόσφατα εγκρίναμε την διαπραγματευτική μας θέση όσον αφορά το κεφάλαιο 8, ανταγωνισμός και λίγες μέρες πριν από αυτό είχαμε και την παραδοσιακή στρογγυλή τράπεζα στην οποία καλέσαμε τους βασικούς εμπλεκομένους που ενδιαφέρονται και περισσότερο στο συγκεκριμένο κεφάλαιο το οποίο είναι σημαντικό όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τη χώρα γενικότερα. Καταγράψαμε λοιπόν σχόλια από όλε τις πλευρές και αυτό μας βοήθησε πολύ στη συζήτηση. Έτσι λοιπόν σφυριλατείται η διαπραγματευτική μας θέση για το κεφάλαιο 8. Αυτό είναι από μόνο του καλό, <laughs> αλλά φυσικά πρέπει να πείσουμε και εσάς, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που έχει επίσης ε, σημασία είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Γι' αυτό έχουμε και μια διακοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία αφιερώνουμε πολλή ενέργεια. Έχουμε συμμετάσχει στην Κόζακ στη Βιέννη, στο Βουκουρέστι και σε άλλες πόλεις. Επίσης, διοργανώσαμε μια περιφερειακή διακοινοβουλευτική σύνοδο, παρόμοια με την Κόζακ δηλαδή, για την δική μας περιοχή, στη δική μας περιοχή. Και αυτό λοιπόν συνέβαλε στο να σημειωθεί πρόοδος στην περιοχή. Όπως ε, είπε και ο βούλγαρος βουλευτής, οι περιφερειακές αυτές κόζακ, αυτές οι μικρές κόζακ, δίνουν την ε, δυνατότητα μεταξύ άλλων να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Τρόικα. Έχουμε και την τοπική Τρόικα, την περιφερειακή Τρόικα, η οποία μας επιτρέπει να συνομιλούμε και να προωθούμε αμοιβαία συμφέροντα. Έχουν γίνει λοιπόν πολλά πράγματα. Χάρη σε όλα αυτά παραμένουμε αισιόδοξοι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία εμφολία ότι το Μαυροβούνιο θα είναι πηγή και αφορμή μόνο καλών ειδήσεων. Όπως πήγε ο κ. Τανό, στην τελευταία διακοινοβουλευτική σύνοδο. Τη επιτροπή μα. Αυτό θα είναι και ένα θετικό μήνυμα για τις άλλες χώρε τη περιοχή στις οποίες ευχόμαστε καλή επιτυχία και τις οποίες βεβαίω θα βοηθήσουμε. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Θα επανέλθω αργότερα αν ε, χρειαστεί κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρυβάκοβιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η άλλη διακριμένη ε, ομιλητέ είπαν ότι είμαι μόνο ένας από πλευρά Είχαμε εξελίξει προ το Βέλτιον, διότι είμαστε στην αρχή τελικά της εφαρμογής των μέτρων για το κάτω δικαίου. Τώρα τι γίνεται το δικαστικό. Εκεί γίνονται διαμαρτυρίες των πολιτών δεν προστατεύονται επαρκώς οι θεσμοί από το πλαίσιο και ο κόσμος θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να πάρει δικαιοσύνη στα χέρια του. Ε, το Σύνταγμά μας θεσπίστηκε το 1792 μετά την Επανάσταση, τη Γαλλική. Τώρα είμαστε στην άνοιξη του Μαυροβουνίου. Δεν έχουμε Επανάσταση. Ακούστηκαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία για προβλήματα. Δεν τα βγάζουν πέρα με τα προβλήματα οι θεσμοί. Έχουμε το Atlas και το Envelope, τα δύο σκάνδαλα. Και βλέπουμε ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα Δυτικά Βαλκάνια, που έχει και Έχει πολιτική οριμότητα το Μαυροβούνιο. Περάσαμε δύσκολες αλλαγές. Με συνένεση στο Κοινοβούλιο θεσπίσαμε την νομοθεσία για το δημοψήφισμα. Μετά το δημοψήφισμα επεξεργαστήκαμε το Σύνταγμα. Το αλλάξαμε το 2013. Και έδωσε περισσότερα δικαιώματα και ανεξαρτησία στο δικαστικό κλάδο το Σύνταγμα και το Σύνταγμα έδωσε μεγαλύτερη προστασία σε αυτούς από ό,τι οποιοδήποτε άλλο Σύνταγμα στην Ευρώπη. Είναι ανεξάρτητοι, έχουν όλα τα εργαλεία, απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και τη δυνατότητα των θεσμών τη βλέπει κανείς όταν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Για το κράτος δικαίου προσπάθησε ξεκίνησα εδώ και 7 χρόνια και στην έκθεση Τάνοκ καλεί τον αρχικό της κυβερνήσεως να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του κάτω δικαίου, την ελευθερία των μέσων ενημέρωση, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματο, οργανωμένο έγκλημα. Και τώρα υπάρχουν πολλέ καταγγελίε για προβλήματα εκεί. Εγώ δεν θέλω να κρίνω, δεν είναι καθήκον μου αυτό. Ήθελα να του πείσω να κάνουν τι αλλαγέ, να γίνουν οι αλλαγέ στο Σύνταγμα. Έγιναν οι αλλαγέ στο Σύνταγμα. Ο λαό βλέπει ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα δεν λειτουργεί, ε, δεν υποδίδει σωστά δικαιοσύνη. Κυνηγάει μόνο τους αντιπολιτευόμενους. Balances are not in, the balance. And uh, distinguished colleagues. συνάδελφοι. Υπάρχουν συμπεράσματα, δηλώσεις που χρειάζονται επικαιροποίηση. Ο κόσμο διαμαρτύρεται ειρηνικά και τα καταστήματα ανοιχτά στι διαμαρτυρίε και στις, ε, στα συλλαλητήρια. Δεν γίνονται πολιτικέ δηλώσει. Απλώ αιτήματα. Έχουν δικαίωμα να έχουν αιτήματα. Η αντιπολίτευση είναι επικοδομητική, πιστεύω. Υπενθυμίζω, 2016 Υιοθετήσαμε λοιπόν την προσωρινή κυβέρνηση που θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Μετά έγινε κρατικό πραξικόπημα. Ε, συνέβησαν πολλά. Μόνο μια διέξοδος απομένει για να χρησιμοποιηθούν. Μέσω προσωρινή κυβερνήσεω να προετοιμαστούν οι εκλογέ. Μέσω υπηρεσιακή κυβερνήσεω. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Έχουμε και πολύ δύσκολα οικονομικά προβλήματα. Χρειάζεται συνένεση και μελλοντικέ εξελίξει αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στο Μαυροβούνιο. Όχι μόνο τι εκλογέ. Οι εκλογέ δεν είναι αποκλειστικό στόχο. Είναι, δεν είναι μόνο στόχο, είναι εργαλείο. ...39 μέλη τη αντιπολιτεύση είπαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές χωρίς υπηρεσιακή κυβέρνηση και είναι η ίδια, το ίδιο ζητάει και ο λαός στο δρόμο. Αυτή είναι μια ευκαιρία για όλους μας. Αν το είχαμε κάνει μια φορά αυτό, το 2016 αν το είχαμε κάνει αυτό, και θα ήταν μια ευκαιρία αν γίνει αυτό για το Μαυροβούνιο. να τα αρνητικά αποτελέσματα να μετατραπούν σε θετικά με τη σωστή προσέγγιση. Και έτσι να συμμορφωθούν με και τις συστάσεις σας. Και η νομοθεσία πραγματικά από εκεί που ήταν η νομοθεσία στα χαρτιά να εφαρμοστεί πραγματικά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η Συμπρόεδρος. Υπάρχουν ε, άλλες παρεμβάσεις. Κάποιος από το πάνελ θα επιθυμούσε να σχολιάσει, μήπως, διαφορετικά. Α, ορίστε. Ο κύριος Μιλόσεβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω όλους. Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλό σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Κρυβόκαπιτς. Απλώς θέλω να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι οι διαμαρτυρίες είναι πολιτικής φύσεως Όλοι το γνωρίζουν το Μαυροβούνιο, όλες οι διαδηλώσεις αυτές. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη που υποστηρίζει μια πλευρά και όχι την άλλη και υποστηρίζει την εξουσία η δικαιοσύνη, υπάρχουν μαρτυρίες. Πόσοι που ήταν σε υψηλές θέσεις, δήμαρχοι κλπ, έχουν ε, διωχθεί. 39 βουλευτές ζητούν η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Όσον αφορά το Δημοκρατικό Κόμμα των Σοσιαλιστών και τα μέλη του συνασπισμού, είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε τα πάντα. Αλλά συμφωνία να συζητήσουμε πρώτα τον εκλογικό νόμο. Όμως κάποιοι βουλευτές έφυγαν από το Κοινοβούλιο και δεν μας επέτρεψαν να συζητήσουμε σωστά το θέμα. Κάποιοι άλλοι βουλευτέ βγήκαν στου δρόμου και είναι στου δρόμου. Και είναι κακή εμπειρία αυτή για μα, Την περασμένη φορά Είχαμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, κυβέρνηση εμπιστοσύνη, όμω μετά τι εκλογέ που διεξήχθησαν με αυτή την κυβέρνηση, ξανά είχαν προβλήματα με την αντιπολίτευση όταν αυτή ιτήθηκε και προσπάθησε να βρει άλλε λύσει πέρα από τι εκλογέ και τα αποτελέσματα των εκλογών. Γι' αυτό θέλω να στείλω ένα μήνυμα εδώ. Θέλω να πω ότι είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση. Θέλουμε η συζήτηση αυτή να διεξαχθεί στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε να συζητήσουμε όλε τι εκκρεμότητε σχετικά με το Μαυροβούνιο κυρίως τον εκλογικό νόμο, να προσπαθήσουμε να συντάξουμε σωστό εκλογικό νόμο, αλλά μπορούμε να βγάλουμε ό,τι αποτελεί εμπόδιο και να βελτιώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Πιστεύουμε όλοι στο Μαυροβούνιο έχουμε αυτή τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο και μετά από αυτό να διεξαχθούν εκλογές που θα αναγνωρίζουν τα, όλοι τα αποτελέσματα. Αυτό είναι προς όφελος όλων και για την εξουσία και για όλους τους πολίτες. Αναφέρθηκαν υποθέσεις, υπόθεση φάκελος, Φερρυπίν. Οι σχετικές αρχές κινήθηκαν εντός των εξουσιών. Η διαδικασία ακολουθείται, έχουν ε, κατατεθεί ε, ποινικέ διώξεις και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Ποτέ δεν είπαμε ότι θέλουμε να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Σε σχέση με αυτά που είπε και ο Σκριβοκάπιτς, θεωρούμε ότι οι θεσμοί πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει και οι ένοχοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Και η υπηρεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς ήδη το, σοσιαλ... το Δημοκρατικό Κόμμα των Σοσιαλιστών το τιμώρησε με κυρώσει και τα χρήματα κατατέθησαν στον κρατικό προπολογισμό. Ε, έγιναν σύμφωνα με την νομοθεσία του Μαυροβουνίου. Αν αυτό δεν αρκεί και δεν είναι καλό ο νόμο, α κάνουμε τι δύο αλλαγέ ε, μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπόχτα. Να συμφωνήσω και να διαφωνήσω. Συμφωνώ, οι διαμαρτυρίε είναι πολιτικέ. Αυτά συμβαίνουν παντού, αλλά οι πολίτε εν τέλει είναι στο κέντρο. Οι διαπραγματεύσει είναι σαφώς, έχουν σαφώ πολιτικά κίνητρα. Περί αυτού πρόκειται. Οι πολίτε θέλουν να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Βλέπουν τους θεσμούς να μην λειτουργούν. Και οι πολίτες αυτό φωνάζουν. Και το δεύτερο. Το θέμα είναι να είμαστε ψύχρεμοι τις ημέρες των εκλογών. Για το καλό κοινό. Αλλά αυτά που έγιναν στις εκλογές δεν τα είδα ούτε στη Ρωσία, ούτε στο Τατζικιστάν, ούτε στο Ουσμπεκιστάν. Για να μην αναφέρω και άλλε χώρε. Και πιστεύω ότι οι εκλογέ ήταν εντάξει. Τέλο πάντων, α το ξεχάσουμε αυτό. Πάμε παρακάτω. Να κοιτάξουμε να κάνουμε σωστά τι επόμενε εκλογέ. Και κλείνω λέγοντα ότι η αντιπολίτευση αυτή τη φορά δεν θα συζητήσει χωρίς αρχικές εγγυήσεις. Το κάναμε το 2015, το κάναμε το 2016. Αυτή τη φορά. Πρώτα θα συμμετάσχουμε στη συζήτηση και θα εξασφαλίσουμε διάφορε ε, εγγύσει στη συνέχεια. Πρώτα θα γίνουμε μέλη τη κυβέρνηση, η κυβέρνηση και μετά θα δημιουργήσουμε τι εγγύησει. Παρακαλώ. Σκρέλα. Oh, Παρακαλώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ κατά πρώτον. Ευχαριστώ όλους που περιέγραψαν την πραγματικότητα στο Μαυροβούνιο. Και είναι αλήθεια ότι κάνουμε βήματα προς τα εμπρός, Γινόμαστε ένα σύγχρονο κράτος, ένα ενεπτυγμένο κράτος. Ευχαριστώ και για το ότι αναφερθήκατε στα επόμενα βήματα. Είπατε μερικοί από εσά ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα στον επόμενο Ιούνιο που θα ξανασυνηθούμε εμεί ω Διακοινοβουλευτική Επιτροπή. Ναι. Πρέπει να έρθουμε πιο κοντά σε αυτό που επιδιώκουμε όλοι μας. Αυτό λέω προς τους συμπροέδρους και τους άλλους παρευρισκόμενους εδώ σήμερα. Προσωπικώς ανησυχώ, όχι για έναν πολιτικό, αλλά για κάποιον που κυβέρνησε τη χώρα 18 χρόνια, όχι 18 μέρες, 18 εβδομάδες, 18 μήνες και ανακοίνωσε την μαυροβουνιακή άνοιξη. Ε, ανησυχώ όταν ακούω τέτοια. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε για να κοιμηθώ κι εγώ ήρεμα το βράδυ. Μου θυμίζουν όλα αυτά αραβική άνοιξη σε ένα σωρό χώρε. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Συγγνώμη. Αυτές οι άνοιξει μόνο κακά πράγματα έφεραν. Και κακά θα φέρουν και στο Μαυροβούνιο. Ο κύριος Κρυβοκάπης τα είπε με το δικό μου τρόπο, είπε ε, ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη και όταν δεν λειτουργεί λέει η δικαιοσύνη, οι πολίτες παίρνουν το νόμο στα χέρια τους. Συγγνώμη, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώνουμε και την ίδια στιγμή κάποιοι να ισχυρίζονται ότι η χώρα δεν πάει καλά, η δικαιοσύνη δεν πάει καλά. Όλοι είπατε ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο στι διαπραγματεύσει. Το σημείωσα. Ότι ήδη βλέπουμε φω στο τέλο τη χειράγγα και ούτω καθεξή. Άρα δεν μπορεί κάποιο να λέει ότι χρειαζόμαστε, κύριε κάποιο μια άνοιξη, μια μαυροβουνιακή άνοιξη. Δεν θέλουμε να δούμε του πολίτε να παίρνουν το νόμο στα χέρια του. Τι θα γίνει Μπορείτε να φανταστείτε μια χώρα όπου οι πολίτε παίρνουν τον νόμο στα χέρια του. Αυτά δεν έγιναν ποτέ. Δεν έγιναν ούτε την εποχή του Χριστού. Ακόμα και τότε υπήρχε δικαιοσύνη, υπήρχαν εισαγγελεί, υπήρχαν δικαστέ. Δεν μπορεί ο καθένα να παίρνει λοιπόν τον νόμο στα χέρια του. Γιατί κάποιοι αντί για τον Χριστό θα επιλέξουν τον Βαραβά. Ε, δεν είναι καθόλου προφανέ το αποτέλεσμα τι γίνεται όταν οι πολίτε παίρνουν το νόμο στα χέρια του. Τώρα, για τις υποθέσεις Άτλας ε, κλπ. Δεν υπάρχει υποθεσία Atlas υπάρχει μια περιοχή στην οποία κάποιος ο οποίος έχασε την επιχείρησή του προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σκάνδαλο, να κατασκευάσει ένα σκάνδαλο. Δεν λέω για την υπόθεση Φάκλος, λέω για την Atlas, έτσι. Η Atlas δεν υπάρχει. Κάποιοι προσπαθούν να κατασκευάσουν την υποτιθεμένη υπόθεση Atlas. Κάποιοι χρησιμοποίησαν ακόμη και φοιτητέ για να περιγράψουν τους εαυτούς τους ως θύματα. Όπω είπε και ο κ. Κρυβοκάπετς, είχαμε διαμαρτυρίες, είχαμε ειρηνικές διαμαρτυρίες. Είναι αυτοί οι οποίοι έχασαν τις δουλειές τους εξαιτίας αυτού του ανθρώπου, ε, είναι φοιτητέ που έχασαν τις θέσεις τους εξαιτία του ίδιου ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο υποστηρίζουν τον Κνέζεβιτς, αλλά δεν κατεβαίνουν στον δρόμο για να τον υποστηρίξουν. Λοιπόν, πολιτικά κίνητρα και εδώ. Φυσικά μπορούμε να βελτιώσουμε το κλίμα, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Κανείς δεν είναι τέλειος άλλωστε, καμία χώρα δεν είναι τέλεια. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα νομοθετήσουμε στον δρόμο και η δικαιοσύνη μπορεί να βελτιωθεί, αλλά δεν μπορεί να βελτιωθεί με διαδηλώσει στους δρόμους. Επίσης, η κρατική ραδιοτηλεόραση. Και αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Αλλά δεν θα γίνουν όλα αυτά με φωνασκίες στα πεζοδρόμια. Αυτά γίνονται μέσω των θεσμών, μέσω των δημοκρατικών θεσμών, μέσω λειτουργικών δημοκρατικών θεσμών. Σε κάποιου θα αρέσουν, σε κάποιου δεν θα αρέσουν, αλλά έτσι γίνονται τα πράγματα στις δημοκρατίες. Ευχαριστώ. Βλέπω έτσι μια πολύ ζωηρή συζήτηση. Να δώσω τον λόγο στον κύριο... Στον Τόμα και μετά στον κύριο Σκυβάκοβιτς. Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά. Ξέρετε, όπω όλε τι ευρωπαϊκές χώρες, η πολιτική κατάσταση δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Το ίδιο ισχύει και για το Μαυροβούνιο. Το σίγουρο είναι ότι το Μαυροβούνιο είναι μπροστά σε σχέση με τι γειτονικέ χώρε. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και προβλήματα. Ότι δεν υπάρχουν προβληματικέ καταστάσει. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση εδώ. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, άσπρο ή μαύρο. Και τα δύο ισχύουν ταυτόχρονα. Πολύ εύκολα. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για την υπόθεση φάκελο, envelope, αλλά υπάρχουν ερωτηματικά, ξέρετε. Τι γίνεται με τον ε, υποδιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας όταν ο διοικητής λέει ότι μία απόφαση των του δικαστηρίου δεν μπορεί να κυρώσει η απόφαση της Βουλής εδώ κάτι δεν πάει καλά. Αυτό δεν είναι μια λειτουργική δημοκρατία. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, γιατί δεν άκουσα κάποιον να το λέει αυτό που σας είπαμε με αυτά τα λόγια, αλλά μου μεταφέρθηκε. Αλλά Σίγουρα πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν στο νομικό πλαίσιο, πολλά μπορούν να γίνουν στην πάταξη της διαφθοράς, ιδιαίτερα σε πολύ ψηλό επίπεδο, εάν και εφόσον συμβαίνει. Και άλλο ένα πράγμα, για να μην είμαι μακρηγορώ. Ναι, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να διαμαρτύρονται αν θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Και αυτή τη στιγμή, και τι παιδιά δεν πάνε στο σχολείο, βγαίνουν ε, έξω και φωνάζουν για το κλίμα. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Και καλό είναι που βγαίνουν τα παιδιά και φωνάζουν για τη μεταβολή του κλίματος. Είναι μια πολιτική διαδικασία. Μιλούν οι μεν με του δε. Καλό είναι αυτό. Και όλα αυτά είναι μέρος και μιας δημοκρατικής εκπαίδευση που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας. Πολλές φορές υπερβάλλουμε, αλλά έχουν το δικαίωμα, επαναλαμβάνω, να διαδηλώνουν. Καλό είναι όλο αυτό. Και είναι εν τέλει το δικαίωμα των πολιτών να ζητήσουν να επιταχυνθούν οι εκλογές. Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εκλογέ νωρίτερα, με την προπόθεση ότι υπάρχει φυσικά η σχετική πλειοψηφία. Τα μεγάλα κόμματα, οι κύριε πολιτικέ δυνάμει δεν έχουν τίποτα να φοβούνται από τι επερχόμενε εκλογέ. Είναι και αυτό κομμάτι τη δημοκρατική διαδικασία. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι καλό που συμβαίνουν. Είναι δημοκρατικέ διαδικασίε, ακόμη και αν καμιά φορά μα μας ανησυχούν οι φωνασκίε και οι διαδηλώσει στου δρόμου. Η δημοκρατία έχει και αυτά. Το πιο σημαντικό που έχουμε στα χέρια μα είναι ακριβώ η δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Στάνισεκ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε κάτι δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί ε, τελεσίγραφα για την εξαγωγή εκλογών. Ακούσαμε κάποιον που, ζη, που είπε ότι χρειαζόμαστε υπηρεσιακή κυβέρνηση και μετά να συνομιλήσουμε. Πρέπει να θετήσουμε νομοθεσία, είπε. Στην νομοθεσία δεν έχουμε μόνο καλά πράγματα. Αν τα είχαμε μόνο καλά πράγματα, θα ήμασταν μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Πρέπει να θετηθούν νόμοι στο Κοινοβούλιο και όχι αλλού. Οι κύριοι της αντιπολίτευσης θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλη η αντιπολίτευση του Μαυροφουνίου υποστηρίζει κάποιον που έχει τελή υποδίωξη και υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του και πρέπει να απαντήσει στο δικαστικό κλάδο του Μαυροβουνίου. Και όλα τα 29 μέλη της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν αυτό που κρύβεται σε άλλη χώρα και υπάρχει ένταλμα σύλληψης του διεθνές. και υποστηρίζεται από κάποιου ΜΚΟ και από κάποια ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση. Έχει δημιουργηθεί μέτωπο να τον προστατεύσει και να μην δικαστεί στο Μαυροβούνιο. Και σκοπό των διαμαρτυριών είναι να σώσουν το κεφάλι αυτού του ζάπλου του ανθρώπου. Είναι πολιτικέ διαμαρτυρίε αυτέ, διαδηλώσει, που στηρίζονται από την αντιπολίτευση, κάποια ΜΜΕ και κάποιες ΜΚΟ και συνάδελφοί μας από το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Ε, είναι, δεν είναι κάτι αληθινό, είναι μια βιτρίνα αυτή. Έχουν το δικαίωμα πράγματι να διαμαρτύρονται οι πολίτες. Είναι ειρηνικέ διαμαρτυρίες. Δεν μπορεί να ζητά κανείς όμως παρέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, και του ανώτατου κρατικού δικαστή. Αυτό είναι επίθεση κατά του κράτους. Δεν είναι κανονικές συνθήκες που ισχύουν σε κανονικές δημοκρατικές κοινωνίες. Δεν μπορεί να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών έτσι. Ε, πέρσι μεγάλωσε, αυξήθηκε σημαντικά η οικονομία μας με τον ταχύτερο ε, ρυθμό, 5% η αύξηση του ΑΕΠ. Το Μαυροβούνιο δεν απειλείται οικονομικά, απειλείται από άλλη πλευρά όμως όπου οι πολιτικοί υποστηρίζουν κάποιον που είναι φυγάς από τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Προτείνω να κλείσουμε αυτό το θέμα. Σίγουρα συνέχεια θα αναδύονται αυτά τα σημεία στη συζήτηση. Σημείο 4 τώρα. Δραστηριότητε Επιτροπή για περαιτέρω μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου και άλλων νόμων. Ούζο Ράντο, εκ μέλου του Κοινοβουλίου, έχει το λόγο πρώτος εκ μέρου του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα. Η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου και τη σχετική διαδικασία στο Μαυροβούνιο είναι μακροχρόνιο θέμα. Μετά τις εκλογές του 2016 δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας στο Κοινοβούλιο και μετά τις εκλογές διεξήχθησαν τοπικές εκλογές και προεδρικές, δημοτικές και προεδρικές. Υπήρξαν αμφισβητήσεις για την εκλογική διαδικασία στο Μαυροβούνιο. Υπάρχουν θέματα που αναφέρονται από τον ΟΑΣΕ και από τους Ευρωπαίους παρατηρητές. Κάποια προβλήματα είναι τεχνικής φύσεως. Κάποιες αλλαγές απαιτούν πλειοψηφία δύο τρίτων, όπως η αλλαγή του συντάγματος. Όλα αυτά είναι στο παρελθόν. Τέλος Οκτωβρίου του 2018 μια νέα προσωρινή επιτροπή συστάθηκε για τον εκλογικό νόμο, για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Μόνο λίγα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην προσωρινή αυτή επιτροπή. Οι δημοκράτες και ούρα το, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στην προσωρινή επιτροπή. Αποφάσισαν να δημιουργήσουν δικό τους βήμα με συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και άλλων πολιτικών παραγόντων, μελών του Κοινοβουλίου και αυτή το εναλλακτικό βήμα, ο φορέας να καταλήξει σε δική του πρόταση για την εκλογική ε, αναθεώρηση. Η επίσημη προσωρινή επιτροπή που δημιουργήθηκε, συστάθηκε από το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου αποτελείται από ίσον αριθμό μελών, μελών της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου και της Αντιπολίτευσης. Με δύο μέλη από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τρεις εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Και προθεσμία για αποβολή πρότασης για μεταρρύθμιση της νομοθεσίας είναι 30 Σεπτεμβρίου του 2019. Πριν ένα χρόνο πριν τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Και υπήρχαν και διάφορε αξιώσει να μην αλλάξει εκλογικό νόμο πριν τη διεξαγωγή των εκλογών. Φιλόδοξο το σχέδιο. Η σύνθεση τη προσωρινή επιτροπή είναι καλή. Έχει 7 ομάδε εργασία που συστάθηκαν με τα ίδια βασικά θέματα, ασχολούνται. Να τονίσω κάποια θέματα μόνο. Το Δικαστικό Συμβούλιο, η νομοθεσία για το δημόσιο σταθμό RTSCG, η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης, μετά όμως από το σχηματισμό της Επιτροπής, λόγω νέων πολιτικών εξελίξεων και αναταράξεων στο πολιτικό τοπίο του Μαυροβουνίου, το Δημοκρατικό Μέτωπο σταμάτησε τη συμμετοχή στην προσωρινή επιτροπή και τώρα η διαδικασία έχει αποτελματωθεί. Και δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι η μελλοντική εξέλιξη. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα και στην προηγούμενη συζήτηση πριν από λίγο. Ε, πίζω ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου με άλλα λόγια, μαζί με άλλους εμπλεκόμενους, δηλαδή τα μέλη της αντιπολιτεύσεως, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών και το κοινό εν γέννη, θα βρουν μια διέξοδο. Πώς να συνεδριάσουν και να συζητήσουν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία για την εκλογική διαδικασία, ούτως ώστε οι νέε κοινοβουλευτικέ εκλογές το 2020 να διεξαχθούν σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία να μην υπάρχουν προβλήματα, να διεξαχθούν οι εκλογές σύμφωνα με τις δημοκρατικές ε, προδιαγραφές. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου του Κοινοβουλίου του Μαυροβούνιου, η κυρία Σκυποβάνοβιτ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας χαιρετίζω και επιτρέψτε μου να σας πω λίγα πράγματα για πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την προσωρινή κοινοβουλευτική επιτροπή και τις δραστηριότητές της. Θα παραλάβω ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση της εκλογική νομοθεσίας είναι μια ισομερής επιτροπή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. σκοπός της είναι να βελτιώσει τη σχετική νομοθεσία, το εκλογικό κλίμα αλλά και τις διαδικασίες. Έχει συγκεκριμένες δραστηριότητες και φυσικά συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Η Επιτροπή αυτή έχει πεπερασμένο χρόνο διάρκειας Λόγω των τελευταίων εξελίξεων, κάποια κόμματα αποφάσισαν να αποχωρήσουν όμως από την Επιτροπή αυτή. Κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάποια κόμματα όμως παρέμειναν και συμμετείχαν στη διαδικασία. Δυστυχώ η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή σαμποτάρει τα πάντα, όχι μόνο την Επιτροπή αυτή, αλλά και τις ίδιες τι ε, συνόδους του Κοινοβουλίου μας. με την εξαίρεση των διεθνών μας δραστηριοτήτων. Εκεί συμμετέχουν. Μετά, οι διαμαρτυρίες λένε οι άλλοι ότι δεν έχουν πολιτικά κίνητρα και όμως έχουν. Ίσα ίσα, κάθε φορά στις πρώτες θέσεις βλέπει κανείς τους εκπροσώπους αυτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εν πάση περιπτώσει, η σχετική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την ε, μεταρρύθμιση της εκλογικής νομοθεσίας συνεχίζει να λειτουργεί, προχωρά. Με ή χωρίς την αντιπολίτευση. Υπάρχουν ομάδες εργασίες, εργασίες οι οποίες ασχολούνται κάθε μία με διαφορετικές πτυχές της σχετικής νομοθεσίας. Τον Σεπτέμβριο, παρά την άρνηση να συμμετάσχουν Βουλευτέ τη αντιπολίτευση. όλες οι ομάδες εργασία συνεδρίασαν, συμμετείχαν πανεπιστημιακοί, μικίο αποφασίστηκε συγκεκριμένη μέθοδος εργασίας για όλες τις ομάδες εργασίας. Έχουμε και μια σχετική γραμματεία, μια γραμματεία αυτής της Επιτροπής, η οποία αναλύει το νομικό πλαίσιο και υποστηρίζει τις επιμέρους ομάδες εργασίας. Μας βοήθησε επίσης ο ΑΣΕ ήταν ε, εδώ, δηλαδή στο Μαυροβούνιο ο ασε το 2016. Συμμετέχουν επίσης και άλλοι διεθνείς οργανισμοί με εμπειρογνωμοσύνη, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε πού χρειαζόμαστε ακριβώ εμπειρογνωμοσύνη για να προχωρήσουμε προ τα εμπρό. Αυτή τη στιγμή, μετά από όλα αυτά, υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, ξέρουμε με ποιου εμπειρογνώμονε θα δουλέψουμε Υπάρχει μια πλατφόρμα εκπαίδευση μεταξύ άλλων του προσωπικού μα, του προσωπικού της γραμματείας. Ε, θα εκπαιδεύσουμε τους ίδιου τους βουλευτέ. Προχωρούμε βλέπετε και σε αυτόν τον τομέα. Επίσης θα διευκολύνουμε το κοινό να συμμετάσχει. Θα πάμε επίσης στην Ιστονία και στην Κροατία. Θα στείλουμε εκεί λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους, κρατικούς λειτουργούς για να μάθουν. Και θα χρησιμοποιήσουμε επίσης και βοήθεια από τις γειτονικές χώρες για να δημιουργήσουμε ένα κοινοβουλευτικό φόρουμ, για να συζητήσουμε ακριβώς την εκλογική διαδικασία. Σίγουρα έχουμε να μάθουμε κάτι από την ε, εμπειρία των γειτόνων μας. Λειτουργεί λοιπόν αυτή η Επιτροπή με μικρή, όπω είπα, με πανεπιστημιακούς και άλλους. Επίσης, έγινε και μια σύσκεψη του ΟΑΣΕ με τα μέλη τη γραμματεία μας, με τα μέλη τη γραμματεία τη Επιτροπής, στο Μαυροβούνιο, με αντικείμενο την διαβούλευση για την κρατική τηλεόραση, την κρατική ραδιοτηλεόραση. ΑΣΕ μας βοηθάει σε αυτήν την διαδικασία. Θα σε έγινε και μια ομιλία από εμπειρογνώμονα από τη Σλοβακία. Το κοινό ήταν ε, η γραμματεία και άλλοι εμπειρογνώμονες. Με βάση όλα αυτά που σας περιγράφω, θέλω να πω ότι αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί διεκπαιριώνει μελέτες, έρευνες. Και φυσικά τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν και στην αντιπολίτευση. Ελπίζω να συμπερταχθούν στην προσπάθεια αυτή. Δεν θέλουμε νόμους μόνο για εμάς βεβαίως. Ο ρόλος αυτής της Επιτροπής είναι πολύ σημαντικός, ξέρετε. Τον ρόλο αυτόν τον εμπιστεύθηκε η Βουλή μας σε μια Επιτροπή. Πρέπει όλοι να συμμετάσχουμε, όλοι να συνεισφέρουμε. Η Βουλή είναι καλύτερη όταν συμμετέχει και η αντιπολίτευση. Πρέπει όλοι να συζητήσουμε πώς θα βελτιώσουμε το κλίμα, το προεκλογικό κλίμα. Αυτά γίνονται στη Βουλή. Ελπίζω λοιπόν ότι και η αντιπολίτευση θα κάτσει γύρω από το τραπέζι. Έχει συμβεί αυτό μερικές φορές, είχαμε και απουσίες, αλλά Ελπίζω ότι θα συνειδητοποιήσουν ότι ο διάλογος γίνεται στη Βουλή. Αυτό είναι και το μήνυμα προς την κοινωνία. Ότι πρέπει όλοι μαζί να τελειώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Αυτό είναι το καθήκον μας. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω κάτι το οποίο εγώ ως μέλος ομάδας εργασίας, είμαι επικεφαλής μάλλον μιας ομάδας εργασίας, η ομάδα μου ασχολείται με τον εκλογικό νόμο. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω την αξία της συνεισφοράς της κοινωνίας των πολιτών που έλαβαν μέρος στην διαδικασία, ήταν στη διάθεσή μας, βοήθησαν πολύ, αλλά ξέρετε αυτό ισχύει και για τους πανεπιστημιακούς και για πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις και εμπειρογνώμονες. Όλοι βοήθησαν Η ανάλυση λοιπόν προχωράει. Καταγράφουμε και τις ανάγκες σε εμπειρονομοσύνη. Όμως να ξέρετε ε, επίσης ότι μας κάλεσαν κιόλας να μιλήσουμε σε διάφορα στρογγυλά τραπέζια. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρετε, από διάφορες ομάδες, από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Λε και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτήν την ε, κοινοβουλευτική επιτροπή. Όλοι περιμένουν να δουν αν κάνουμε καλά τη δουλειά μα. Συμμετέχουν και τα ευρωπαϊκά όργανα. Έχουν καταθέσει τι απόψει του. Γιατί εν τέλει θέλουμε έναν νόμο ο οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί. Δεχθήκαμε και αλλαγέ που πρότειναν ΜΚΟ. Ε, αυτό ήταν και το νόημα της δημόσιας διαβούλευσης. Επίσης κάποιες άλλες πτυχές θα καλυφθούν από άλλους νόμους, για τα μέσα για παράδειγμα. Τροποποιούμε επίσης τον νόμο για την χρηματοδότηση των κομμάτων. Τον νόμο επίσης για τα μέσα. Ε, πολλοί περιμένουν επίσης άλλες αλλαγές, άλλους τομείς. Ε, άτομα με αναπηρίες για παράδειγμα. Για να τροποποιηθούν επίσης κάποιοι νόμοι, σημειώστε ότι χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων. Σε κάθε περίπτωση ο κόσμος περιμένει πολλά από εμάς. Ελπίζω να το καταλάβει αυτό και η αντιπολίτευση. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη. Η ευθύνη μας είναι μεγάλη. Το ξαναλέω, θα ήταν αντιθέτως ανευθυνότητα έναντι των πολιτών μας, έναντι του λαού του Μαυροβουνίου, να επεμπολίσουμε αυτήν την μεγάλη ευθύνη. Συναισθάνομαι λοιπόν την ευθύνη, ε, ελπίζω να τον συνισταθεί και η αντιπολίτευση. Τα μποϊκοτάζ δεν οδηγούν πουθενά. Είναι το δικαίωμα καθενό βεβαίω να μποϊκοτάρει την προσπάθεια, αλλά με τι διαδηλώσει στου δρόμου δεν πάμε μπροστά. Ε, μπορεί κανεί να διαδηλώνει είναι να υποστηρίζει διαδηλωτέ, αλλά ο χρόνο τελειώνει. Ό,τι να κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν ο συνάδελφος Ράντος είπε ότι υπάρχει καταληκτική προθεσμία για τη δουλειά μας. Ελπίζω λοιπόν ότι θα τα καταφέρουμε εντός της προθεσμίας. Να πω εν κατακλείδη ότι έχουμε και τα τεχνικά ζητήματα, την τεχνική της διακυβέρνησης όπως την περιγράψε κάποιος. Προς τούτο χρειάζεται διάλογος. Το 2016 είμαστε μια από τις σπάνιες κυβερνήσεις συνασπισμού. Η αντιπολίτευση ζητούσε να εκπροσωπηθεί δυσανάλογα και σε τοπικό επίπεδο. Τους δώσαμε περισσότερα από ό,τι δικαιούντο, το 2016 αυτά. Και δυστυχώς δεν σεβάστηκαν καν αυτόν τον ειδικό νόμο, τον Lex Specialis, που τους έδωσε υπέρμετρη εξουσία και σε τοπικό επίπεδο. Το θέμα είναι να έχουμε εκλογές βάσει νόμων που δεν θα αμφισβητηθούν ξανά. Πρώτο γεγονός ότι οι εκλογές που έγιναν ήταν απολύτως νόμιμες. Η αντιπολίτευση Απλώ διαμαρτυρήθηκε μόνο εκεί που έχασε. Ήταν καλό ο νόμο ε, εκεί που κέρδιζε, αλλά δεν ήταν καλό εκεί που έχανε. Έτσι λοιπόν άρχισαν να αμφισβητούν το αποτέλεσμα. Τα ζήσαμε αυτά λοιπόν το 2016. Δεν βγάλαμε άκρη. Και τώρα δυστυχώς η αντιπολίτευση για άλλη μια φορά προσπαθεί να καταλάβει την εξουσία χωρίς εκλογές. Αυτά δεν γίνονται. Αυτό είναι παράνομο. Αυτό είναι δυστυχώς. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι θέλει να μιλήσει και ο Σκοβάκοβιτς, αλλά μας τελειώνει ο χρόνος. Ξέρω ότι έχετε κάποια νέα θέση. Να σας δώσω ένα λεπτό και να προχωρήσουμε μετά. Μας λείπει ο χρόνος. Κοιτάξτε, εγώ είμαι μόνο μου και έχω τα δικαιώματα, εκπροσωπώ τα δικαιώματα τη αντιπολίτευση. Υπάρχει η ιστορία τη Προσωπική Επιτροπή του Γιουγκοσλαβία. Επιμένανε στη Γιουγκοσλαβία, κάποιο επέμενε ότι ε, είναι η Ιγκοσλαβία όταν είχαν φύγει τέσσερι δημοκρατίε από την Γιουγκοσλαβία. Ε, το DPS κάνει το ίδιο. Κανεί δεν θέλει να πάει σε αυτή την επιτροπή. Ο κόσμο είναι στου δρόμου έχει πρόταση αντιπολίτευση, α συζητήσουμε την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είδαμε τι έγινε σε εκλογέ παρόλο την υπηρεσιακή κυβέρνηση την προηγούμενη φορά. Είναι τυφλοί, δεν βλέπουν ε, τι γίνεται. Έχετε τα πραγματικά στοιχεία. Αυτός ο οποίος διώκεται πρέπει να έχει την ίδια τύχη και δέχτηκε να πάει στο δικαστήριο. Αυτός που λέει ότι ξεφεύγει. Πώς να μπει στη χώρα όταν δεν υπάρχει σωστός δικαστικός τομέας. Υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία αποδείξεις. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός Μαυροβουνίου και αλλού. Και θα δείτε πώς λειτουργεί η δίκαιοσύνη. Εμάς δεν μας κάνει όμως το σύστημα. Εμείς να κάνουμε τη δουλειά μα θέλουμε, την πολιτική ατμόσφαιρα. Είναι δυνατές οι εκλογέ και υπάρχουν και είναι λειτουργικές οι Είναι δυνατές. Αν θα είναι δίκαιε, είναι άλλο θέμα. Όλα τα άλλα ανήκουν στο δικαστικό κλάδο αν τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά για τον Τουσκοκνέζιτς. Ξέρω και ότι άλλοι θέλουν να μιλήσουν. Η ε, κυρία Μαγκίνες έχει καταφτάσει, είναι μαζί μας και υποψιάζουμε θα μπορέσει να έρθει αργότερα. Για ένα λεπτό. Κοιτάξτε, να κάνω δύο δηλώσεις. Πρώτα απ' όλα δεν συμφωνώ ότι αυτή η Επιτροπή έχει αυτά τα προβλήματα. Αυτή την Παρασκευή συνάντησα δύο εκπροσώπους ΜΚΟ και νομίζω ότι υπάρχει η νομιμότητα να εξεταστεί ο εκλογικός νόμος στο Μαυροβούνιο. Υπάρχει συμμετοχή και της κοινωνίας των πολιτών. Μπορούμε να ξεπεράσουμε τις αρχικές απαιτήσει και μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο και να έχουμε εκλογικό νόμο για τον οποίο θα είμαστε υπερήφανοι και θα αποδεχτεί η αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να εξισώνουμε κάποιον ο οποίος είναι στο ένταλμα σύλληψης της Ιντερπολ με τον πρόεδρο του Μαυροβουνίου. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ότι αυτός είναι νόμιμος και οι θεσμοί δεν είναι νόμιμοι για την αντιπολίτευση. Να κλείσουμε λοιπόν το θέμα αυτό τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου στις 5 πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Μπράγεβης για να προεδρεύσει το επόμενο σημείο. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 5. Βιωσιμότητα των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ε, μεταρρυθμίσεων. Η κυρία Μακίνες, δύσκολη μέρα για όλους μας. Θα είμαι σύντομη. Αν δούμε την έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2018, το Μαυροβούνιο έκανε κάποια πρόοδο και είναι αρκετά έτοιμο όσον αφορά τι μεταρρυθμίσει, τι οικονομικέ και τι δημοσιονομικέ. Η οικονομία αυξάνεται το 2013, βελτιώνεται χωρί διακοπή όσον αφορά το κεφάλαιο 8 ανταγωνισμό. Σύντομα θα είναι το τελευταίο από τα 33 κεφάλαια που θα ανοίξει και αυτό συζητείται στο Συμβούλιο τώρα. Βέβαια πρέπει να κλείσουμε και κεφάλαια εάν δείτε οικονομικό και δημοσιονομικό τομέα δεν έχουν γίνει αρκετές βελτιώσεις. Υπάρχει μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και μεγάλο δημόσιο χρέος, κρατικό χρέος. Αυτά είναι προβλήματα. Υπάρχει, ε, είναι ευάλωτη η οικονομία στις αλλαγές ε, και το δημοσιονομικό δυναμικό είναι χαμηλό και η αδυναμία στο κράτος δικαίου, διαφθορά, η άτυπη οικονομία και η επαχθής νομοθεσία που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Είναι προβλήματα. Το Μαυροβούνιο βεβαίω θέλει να έχει εύρυθμα λειτουργού σε οικονομία τη αγορά. Η, η, σταθερότητα έχει βελτιωθεί στον οικονομικό τομέα, αλλά χρειάζονται και άλλε προσπάθειε στου τομεί αυτού, κυρίω για το μεγάλο κρατικό χρέο, για το κράτο δικαίου οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές διότι επηρεάζουν την οικονομία και όταν υπάρχουν δυναμίες στο κράτος δικαίου όπως η αθέμητος ανταγωνισμός από την άτυπη οικονομία εκεί έχουμε αρνητικό αντίκτυπο στη, στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το Μαυροβούνιο είναι στην 77η θέση από τις 137 χώρες στον κόσμο στην έκθεση του World Economic Forum για την ανταγωνιστικότητα, αλλά υπάρχουν παράγοντες που οδηγούν σε προβλήματα και δυσκολίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις να επιχειρούν. Προσβάσει στην χρηματοδότηση, ε, ανεπαρκείς ε, ε, ε, γραφειοκρατικές δομές στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει αρκετή υποδομή ε, και το εργατικό δυναμικό δεν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες και εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Απαράδεκτα υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων, περίπου το 1 τρίτον των νέων είναι άνεργο Εντάχει να αναφερθώ σε κάποια άλλα σημεία. Καλή πρόοδο έχει επιτευχθεί όσον αφορά το σχέδιο για την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο όσον αφορά οικονομική νομισματική πολιτική. Το Μαυροβούνιο έχει θεσπίσει νομοθεσία που προβλέπει την ανεξαρτησία τη Κεντρική Τράπεζα, αλλά χρειάζεται προσπάθεια τόσο να εξασφαλίζεται αυτή η ανεξαρτησία και να είναι ασφαλή στην πράξη ε, περαιτέρω προσπάθεια χρειάζεται για ευθυγράμμιση με το κεκτημένο, συμμόρφωση με κανόνε Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την πρόληψη προνομιούχα πρόσβαση από το δημόσιο τομέα σε χρηματοπιστωτικού οργανισμού και υπέβαλε η κυβέρνηση την οικονομική μεταρρύθμιση 2018-2020 όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Εν γέννη, οι δυνατότητε των, των δημοσίων αρχών να επιβάλλουν τι διάφορε αναγκαίε μεταρρυθμίσει βελτιώνται σταδιακά γιατί τη φορολόγηση είναι από κάτι και εκεί θα κλείσω. Το Μαυροβούνιο θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα πρέπει να συσχετιστεί με τον <clears throat> ΟΣΑ όσον αφορά αυτό και να συμμετάσχει στο Global Forum για διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών του ΟΣΑ για τα θέματα της φορολογίας. ήμουν σύντομη. Ελπίζω να ήταν μια σύντομη και περιεκτική παρουσίαση. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, κύριε Δελπέρσκα. Πρόεδρε. i naravno gospođi koja je prije govorila što su mi uštedili dodatno vrijeme i naravno na trudu da dodatno objasnim Ok. Da dodatno objasnim Υπήρχε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, έλεγα το εξή όσον αφορά την, τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τις προβλέψεις για την επόμενη τριετία. Όπως είπε και ο κύριος Βουξάνοβιτς, το κεφάλαιο 8 δεν αποτελεί τυπικό θέμα. Η ανταγωνιστικότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό η δική μας ανταγωνιστικότητα θα ενισχύσει αυτήν της Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά και εμείς αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα με αυτά που αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο. Φέτος, πάντως, συμμορφώθηκε το Μαυροβούνιο με συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ξέρετε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν την μεθοδολογία που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν δύο σενάρια μπροστά μας. Το πρώτο είναι το απεσιόδοξο της ε, βραδύτερης ανάπτυξης παρά το γεγονό ότι το Μαυροβούνιο αναπτύχθηκε τελευταία ταχύτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το μέσο όρο της περιοχής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων των διεθνών οργανισμών, το Μαυροβούνιο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό μεταξύ 3,7 που λέει η Κομισιόν και 4,1 που λένε οι δικοί μας οργανισμοί ή και το ΤΑΦ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Οι δύο τελευταίοι πιστεύουν ότι μπορούμε να κρατήσουμε το ρυθμό αυτό μέχρι την ένταξη. Λοιπόν, αν και το είπατε, ναι, χρειαζόμαστε ε, βιώσιμες χρηματοδοτήσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, περιβάλλον φιλικό προς τις επιχειρήσεις. Αυτά τα έχουμε πει. Πρέπει να κάνουμε πράγματα για τις επιχειρήσεις, αυτό είναι βέβαιο. Εκεί δυστυχώ, στη φιλικότητα προς τις επιχειρήσεις, πέσαμε στην παγκόσμια κατάταξη κατά οκτώ θέσεις. Ενδεχομένω η αιτία δεν είναι η επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματο, αλλά άλλες Εξελίξει. Ίσως το ότι κάποιες χώρε έγιναν αυτές καλύτερες και αυτό μας άφησε εμά πίσω. Το θέμα είναι λοιπόν να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Χρειαζόμαστε διαρθρωτικές, όπω είπα, μεταρρυθμίσεις, μείωση των δημοσίων δαπανών. Πρέπει να περικόψουμε τις δημοσίες δαπάνες κατά 5% τουλάχιστον. Και όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, εκεί θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις δαπάνες κατά 10% και αυτό θα οδηγήσει πιστεύω σε ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να πω επίσης ότι το Μαυροβούνιο ζει μεγάλες περιφερειακές ανισότητες. Τα νέα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση αποσκοπούν στην άμβλυνση αυτών των ανισοτήτων υπέρ των λιγότερο ευνημένων περιοχών. Επίσης, προσπαθούμε να επιβάλλουμε συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία. Τα χρέη είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το Μαυροβούνιο κατάφερε να εισπράξει περισσότερου φόρους, να έχει υψηλότερα φορολογικά έσοδα σε σχέση με τις προβλέψεις και αυτό ήταν καλή εξέλιξη. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι επίση ενδιαφέρον είναι το εξή. Στο Μαυροβούνιο ψηφίστηκε νόμος περί οικονομικής ηθαγένειας, ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενος νόμος, με περίπου 200 αιτήσει χορήγησης ηθαγένειας, δηλαδή, με βάση οικονομικά κριτήρια. Το παρακολουθεί το θέμα και η Κομισιόν πολύ προσεκτικά, να ξέρετε. Πάντω ε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να εισφέρει στη χώρα περίπου ένα επιπλέον δισεκατομμύριο. Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, είναι 75% του ΑΕΠ, πολύ ψηλό βέβαια. Το 2017 ήταν 60%. Η αύξηση οφείλεται στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας υπέδειξε πού έπρεπε να επενδύσουμε περισσότερο. Είμαι λοιπόν κεφαλαϊκές επενδύσεις, επενδύσεις σε πάγια, για να μπορέσουμε ακριβώς να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, για να βελτιώσουμε υποδομές, και για να βελτιώσουμε το επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος στο Μαυροβούνιο. Αυτό θα είναι υπέρ του τουρισμού, αλλά και υπέρ της γεωργίας. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα νοοτροπίας. Σύμφωνα με την Eurostat και τις στατιστικές της, η ενέργεια είναι σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα στο Μαυροβούνιο. Θεσπίσαμε βεβαίως μέτρα για να παρακινήσουμε τον πληθυσμό να εργαστεί ως αυτοπασχολουμένος. Επίσης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καταφέραμε πολλά, καταφέραμε πραγματικά 25.000 άνθρωποι να ξεκινήσουν τις δικές τους ατομικές επιχειρήσεις. Πολλοί νέοι, πολλά θύματα της μετάβασης. Όλο και περισσότεροι λοιπόν δραστηριοποιούνται ως αυτοπασχολούμενοι. Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνδράμε στην μείωση της ενεργείας. Ελπίζουμε ότι θα μειώσουμε την ενεργεία κατά 0,9% περαιτέρω. Αυτά το 2019 και ότι θα σταθεροποιήσουμε γενικότερα και την οικονομία με τρόπο αποδεκτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ, κύριε Παγιόβιτ. Κλείνουμε με την εισαγωγή. Οπότε, παίρνουμε στη συζήτηση, αν και ο χρόνο που απομένει είναι ελάχιστο, γιατί οι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να φύγουν για την ψηφοφορία στι 5 το αργότερο. Παρακαλώ. Δεν είχα την ευκαιρία προηγουμένω να πω το εξή. Γενικά νομίζω ότι όλοι είμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου, έτσι δεν είναι. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει. Κάποιοι θέλουν να μας κάνουν λιγότερο ίσους ενώπιον του νόμου και της δικαιοσύνης. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Μαυροβουνίο. Όλοι είναι ίσοι, αλλά κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Αυτά, αυτή είναι και η ιστορία της ανθρωπινής ιστορίας. Δεν θα αναφέρω ονόματα, Τζουγκάνοβιτς, αλλά κύριε Μαγκίνες, ε, πέσαμε 23 θέσεις. 23 θέσεις στην κατάταξη του Heritage Foundation για την ποιότητα της δημοκρατίας. Πριν καν γίνουν όλα αυτά. Τρεις θέσεις πέσαμε και σε άλλε κρατάξει. Ε, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Πέφτουμε παντού. Σε διαφορέ κρατάξεις για ελευθερίες, πολιτικές κλπ. κλπ. Και αυτό έλεγα προηγουμένως ότι χρειαζόμαστε ενότητα. Όχι για πολιτικούς όχι για πολιτικές σκοπιμότητες. Μετά, έπεσαν οι μισθοί κατά 3%. Αυξάνονται οι φόροι. Έχουν ε, πολλαπλησιαστεί επί 7 σε σχέση με την εποχή της ανεξαρτησίας μας. Εξωτερικό εμπόριο, το έλλειμμα είναι γύρω στο 56%. Και γιατί εισπράττουμε τόσο υψηλού φόρου. Γιατί δυστυχώ ε, το κράτο έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η κυβέρνηση δηλαδή. Για του πλούσιου και του φτωχού. Και έχουμε επίση το χαμηλότερο ελάχιστο μισθό στην περιοχή. Το Κόσοβο είναι καλύτερο. Η Μακεδονία καλύτερο. Υψηλότερο ελάχιστο μισθό. Η Βοσνία Η βενζίνη επίση είναι ακριβότερη από οπουδήποτε στην περιοχή το ηλεκτρικό ρεύμα το ίδιο, το ακριβότερο της περιοχής, ε, μια δυσαναλογία απίστευτη. 80.000 άνθρωποι, οι μισοί εργαζόμενοι δηλαδή, οι μισοί υπάλληλοι, παίρνουν μισθό, έχουν μισθό κάτω από 250 ευρώ το μήνα. Και γι' αυτό ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Δεν είναι μόνο αυτά που λέγατε προηγουμένως. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ε, ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους. Η δικαιοσύνη, η πολιτική κατάσταση κλπ. Οι εξήρμοι συνάδελφοι είπαν ότι υπάρχει ένα πελατοκεντρικό σύστημα στην χώρα, ότι υπάρχει διαφθορά. Ναι, υπάρχουν. Ε, και αυτό εξηγεί τις ε, αρνητικές τάσεις. Ναι, αναπτυσσόμεθα με 5%. Αλλά πώς. Και αυτό δεν είναι κάτι που είναι βιώσιμο τα επόμενα χρόνια. Όταν σταματήσουν οι επενδύσεις στους αυτοκινητοδρόμου, τελειώσαμε. Οι μισθοί δεν αυξήθηκαν και δεν θα αυξηθούν. Γιατί έχουμε μεγέθυνση. Δείτε την πραγματική κατάσταση. αυτοί που κατασκευάζουν τους αυτοκινητοδρόμους δεν, δεν πληρώνουν φόρους, αλλά η οικονομική κατάσταση δεν είναι μόνο η αυτοκινητόδρομη Η βενζίνη, όπως είπα, είναι ακριβότερη από οπουδήποτε στην περιοχή. Ο κόσμος πηγαίνει στη Βοσνία για να βάλει βενζίνη. Στη Βοσνία. Όχι στα Αραβικά Εμμυράτα ή τη Σαουδική Αραβία. Στη Βοσνία πηγαίνουν για να βάλουν βενζίνη. Είναι 20% φθηνότερη βενζίνη εκεί από ότι στο Μαυροβούνιο. Κάποιοι κλείνουν τα μάτια, λένε θέλουμε εκλογές, έχουν διπηρετικούς πυράβλους. Το παλιό σύστημα δεν είχε μέλλον, ήταν αναχρονιστικό. Εμείς μπήκαμε σε μια μετάβαση με τρόπο ειρηνικό. Είναι η λύση για να μην ε, περιπέσουμε σε βαθύτερη κρίση. Η κρίση λοιπόν δεν αποσοβήθηκε τα τρία τελευταία χρόνια. Έγινε μάλιστα χειρότερη. Ε, δεν είμαστε στο χειρότερο σημείο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Να ξέρετε, η κρίση θα επιδεινωθεί περαιτέρω. Ελπίζω να υψευστώ, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και όριμοι άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι στο κόμμα του Τζουκάνοβιτς. Και να πω την αλήθεια, υπάρχουν και άνθρωποι στο κόμμα του που θέλουν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει, αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να, κάνουν, να γίνει τίποτα. Αυτό θα δημιουργήσει περισσότερη αστάθεια Ελπίζω ότι κάτι θα γίνει για να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο κοντά στην ένταξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας δώσω το λόγο. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι μιλάμε μόνοι μας. Διότι οι ευρωβουλευτές έχουν φύγει από την αίθουσα για να ψηφίσουν. Λυπάμαι όπου ο κ. Κρυποβάτσης καταχράστηκε του θέματος για να συζητήσει το προηγούμενο θέμα. Αν λέγατε αυτά που είπα σωστά, ποτέ δεν θα βρίσκατε υποστήριξη για τα επιχειρήματά σας. Εγώ αναφέρθηκα σε εντελώς διαφορετικές κατηγορίες. Δεν κατανοείτε και λυπούμε, διότι βάσει αυτών που είπε και ο Σκρέλια και εκείνων που υπενόησε, άλλα ήταν τα εννοήματα. Αυτά που είπα σήμερα ευθυγραμμίζονται με το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης που είναι πλήρως εφαρμοσμένο με τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τη διάγνωση προβλέψεις και συμφωνούμε με αυτούς βάσει αυτού του προγράμματος ότι οι προβλέψεις είναι όπως περιγράφησαν. Γιατί είναι αυτές οι προβολές και οι προβλέψεις δεν τα πάντα ιδεώδη, αλλά πρέπει να μάθουμε και να καταλάβουμε ότι όλα τα βήματα που κάνουμε για καλύτερο κοινωνικό περιβάλλον δεν μπορεί να δημιουργηθεί από, μόνο από τα δικά μας χέρια, αλλά πρέπει με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να συνεργαστούμε που υποστηρίζουν την οικονομία του Μαυροβουνίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βλέποντας τι προβλέψεις για αυτά πρέπει να κάνουμε. Όσον αφορά την, ε, το κόστος τη εργασία, διαφωνώ με κάτι. Ότι δεν υπάρχει καλή βούληση, αλλά θα πρέπει να βρούμε αρκετό περιθώριο στον προπολογισμό για να υποστηρίξουμε ένα υψηλότερο ελάχιστο εισόδημα και να δούμε κατά πόσο αυτό θα είναι απορριθαρρυντικό για το σύστημα κοινωνική πρόνοιας. Δεύτερον, να δούμε το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο μπορούμε να αυξήσουμε την το ελάχιστο μισθό και να μην αποσταθεροποιήσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Γιατί με ψηλέ αμοιβέ θα έχουν ακόμα ψηλότερε αμοιβέ και αυτοί με ελάχιστο εισόδημα δεν θα ωφεληθούν πολύ από την αύξηση του ελάχιστου μισθού. Θα πρέπει να φροντίσουμε να ακολουθήσουμε σωστή θέση όσον αφορά την αύξηση του ελάχιστου μισθού, όσον αφορά το επενδυτικό περιβάλλον. Ειλικρινά ελπίζω ότι οι προβλέψεις για το 3,7% που είναι πιο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης αποδεικνύει αν αποδειχτεί αυτή η ανάπτυξη, αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης και οι δικές μου και οι δικές σας αμφιβολίες θα εξαλειφθούν αν όλοι αυτοί οι στόχοι επιτευχθούν. Ευχαριστώ. Ο κ. Χάιντλάιτνερ έχει το λόγο. Uh, uh, Συζητάμε την οικονομία. για τη μεταρρυθμιστική διαδικασία και τα διάφορα σχόλια των ομιλητών. Έχω το συνέστημα καμιά φορά ότι το Μαυροβούνιο εστιάζεται πολύ στις μεγάλες επενδύσεις. Τα μεγάλα έργα υποδομών για οικονομική ανάπτυξη και δεν συγκεντρώνεται αρκετά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη δημιουργία επιχειρήσεων. Όταν μιλάμε με τους διάφορους οικονομικούς φορείς, οι εκπρόσωποι των μεγάλων εταιριών διαμαρτύρονται κυρίως για την άτυπη οικονομία. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι στο σύστημα και διαμαρτύρονται για αυτές που δεν είναι στο σύστημα, διότι δεν είναι ισότιμες οι συνθήκες ανταγωνισμού. Και θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτά τα θέματα. Να εξασφαλιστεί ότι οι περισσότερες εταιρείε συμμετέχουν στο σύστημα και αυτοί που είναι στο σύστημα να μπορούν να λειτουργούν σύμφωνα με τους ίδιους όρους. Και έτσι θα ξεκλειδωθεί ένα μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης στο Μαυροβούνιο. Τη τη οικονομίας του Μαυροβουνίου. Από εκεί μπορεί να προέρθει ανάπτυξη. Και αξιολογώντα το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης για αυτό το χρόνο, εστιάζεται κυρίως στη μείωση της άτυπης οικονομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Πρέγεβιτς. smo kroz analizu koju smo interno radili barem mi u parlamentu u crnoj gori imate šest hiljada firmi koji imaju samo jednog zaposlenog λοιπόν η κυρία Πρέγεβιτς το Πρέγεβιτς δεν συμπεριλάβανε κάποια στοιχεία έχουμε 6.000 μικρές εταιρείες στο Μαυροβούνιο με μόνο έναν εργαζόμενο στη μεταποίηση τραφήμων. Υπάρχει, υπάρχουν εταιρείε με έναν φορολογούμενο καταχωρημένο. Ένα είναι καταχωρημένο σε κάποιε επιχειρήσει και 20 δεν είναι. Σε ξενοδοχείο 10 καταχωρημένοι επίσημα εργαζόμενοι και άλλοι δεν είναι. Άρα χρειάζεται έλεγχο. Εκεί πρέπει να βασιστούμε στου ελέγχου. Να εξαλειφθούν αυτέ οι παρατυπίε για να ξεκινήσουν οι κύκλοι που αναφέρατε. Και να ελέγξουμε τι μικρέ εταιρείε τις εταιρείε που θέτουν νέες έννοιες, όπως αυτή από την Τουρκία που έρχονται στο Μαυροβούνιο. Είναι μια νέα εξέλιξη στην οικονομία του Μαυροβουνίου. Δεν θέλουμε να κάνουμε σφάλματα που ήδη έχουν εντοπιστεί προηγουμένως στο Μαυροβούνιο. Αν υπάρχει σωστός έλεγχος, θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αν έχουμε θετικά αποτελέσματα, θα είναι καλά παραδείγματα για την καταχώρηση νέων μικρομεσών επιχειρήσεων και να εφαρμόσουμε και τις αρχές που Ευχαριστώ. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 6 και θα συνεχίσουμε στις 6.